ξεκινώντας να δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στον πρόεδρο Πέτεριν, ο οποίος τιμά κάθε χρόνο τη διάσκεψή μας με την παρουσία του. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητή μου Άννα Σαπόσκα, αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητή Μαργκότ Βαλστρούμ, κύριε Επίτροπε Βλαντιμίρ Σπίτλα, κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια όλος εξαίρετη ευκαιρία σήμερα να συναντηθούμε και γι' αυτό απευθύνω ιδιαίτερα σημαντικό για μένα χαιρετισμό. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων σα των κοινοβουλίων μας, ε, στην αίθουσα τη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων τη γυναίκα και της ε, ίσης των γυναικών ε, είχε την τιμή να με προσκα... μου έκανε τιμή να με προσκαλέσει για να εορτάσω μαζί τη την ε, Διεθνή ημέρα τη γυναίκα και την ευκαιρία αυτή τη ε, εκκίνησης των εργασιών τη διάσκεψης για την γυναίκα στις ευρωεκλογές. Σα ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα και για την πρωτοβουλία σας, ιδιαίτερα την ε, κυρία Πρόεδρο Αναζαμπόρσκα, η οποία ε, πάντοτε με τόσο ενδιαφέρον αγωνίζεται για τα θέματα αυτά. Βρισκόμαστε μερικούς μήνες μόλις πριν από τις ευρωεκλογές. 90 ε, μέρες περίπου θα έχουμε 375 εκατομμύρια πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών που θα έχουν την ευκαιρία τον Ιούνιο να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για τα επόμενα πέντε χρόνια. Είναι λοιπόν η στιγμή αυτή η καταλληλότερη για να συζητήσουμε και τον ρόλο που διαδραματίζει η γυναίκα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, να τον αναλύσουμε, να τον αναπτύξουμε. Και τώρα όσο μιλάω βλέπω ότι μάλλον έφτασε κάποιο αεροπλάνο από κάποιο μέρος της Ευρώπης γιατί ε, αμέσως εκδηλώνεται ξαφνικά αθρώα ε, έλευση ακροατών. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και τα εθνικά κοινοβούλια ε, ιδιαίτερα στρατεύεται στην στον αγώνα για την δημοκρατική εξέλιξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα των κοινωνιών μας. Μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ αρχής ήταν η ε, αναγνώριση του ρόλου της κοινωνίας στην, της γυναίκας στην κοινωνία και η εξασφάλιση όρων εργασίας ε, ε, και ζωής στην κοινωνία των πολιτών και την πολιτική ισότιμων και για τη γυναίκα. Αποτελεί λοιπόν η εξίσωση, η ισότιμη μεταχείριση των ε, φύλων για την Ευρωπαϊκή Ένωση κύριο αγώνα. Βάση της ισότιμης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών αποτέλεσε, έστω και με κάποιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, ήδη η συνθήκη της Ρώμης του 1957, όπου στο πεδίο εφαρμογής της αναφέρεται και διατυπώνεται η ισότιμη μεταχείριση των φύλων, όπου βέβαια ήδη, ε, η οποία ήδη βρίσκει την έκφρασή της και στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας σήμερα, ύστερα από προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής, λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα έχουμε ε, σημειώσει ένα πολύ σημαντικό βήμα προόδου στην ισότητα μεταχείριση των φύλων, όταν θα εγκριθεί και θα τεθεί εν τέλει μετά την κύρωσή της σε ισχύ η ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν βρίσκεται στον, ε, στην πρώτη γραμμή των ε, αγώνων μας. Το 1979 γίνεται γυναίκα η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγόμενου κοινοβουλίου που πρώτη φορά εκλέχθηκε με άμεση ψηφοφορία το 1979 και η πρώτη πρόεδρος ήταν γυναίκα η κυρία Σιμών Βέιλ την οποία μάλιστα προσκαλέσαμε και επίσης έχουμε και την μεγάλη μορφή της Λουίζε Βάης, εκείνης η οποία ανακήρυξε πρώτη την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκείνου το 1979 στην οποία είχα την τιμή να είμαι και εγώ παρόν, λόγω τη ηλικία σα, γιατί πάντοτε το ξεκίναω πρεσβύτερο των βουλευτών την τακτική συνέλευση του Κοινοβουλίου. Και ε, όπω είπα λοιπόν, είχα την τιμή να είμαι εγώ παρόν και μπορώ να σα πω χωρίς έξω από το κείμενό μου ότι γνωρίζω πολύ καλά το σύστημα που ακολουθούσε το κόμμα της κυρίας ε, Βάης είχε α, στηριχθεί στο σύστημα του γουλμό, όπως το λέγανε στη Γαλλία, δηλαδή την ε, ε, εναλλάξ προβολή ανδρών ή γυναικών κατά περίπτωση στους ηγετικούς θόκους του κόμματος. Η Λουίς Βάης λοιπόν εκείνη ήταν η μορφή η οποία μπόρεσε χάρη στην εναλλαγή αυτή να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, στην ηγεσία του κόμματό τη, στην ε, επόμενη χρονιά που θα έπρεπε να γίνει η εναλλαγή, δεν υποχώρησε και μπόρεσε χάρη στη δύναμη του χαρακτήρα τη και την προσωπικότητά τη να επιβληθεί και να ε, χαρακτηρίσει με την παρουσία τη ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 1979 λοιπόν εκλέγεται, αναφέρομαι πάλι στο πρόσωπο της Σιμών Βέιλ, η πρώτη μας πρόεδρος, η πρώτη εκλεγόμενη, εκλεγμένη πρόεδρος, αν και θα πρέπει να σας πω ότι ήταν το Αυστριακό Κοινοβούλιο εκείνο το οποίο έκανε την πρωτιά το 1927 όπως έμαθα προετοιμαζόμενος για τη σημερινή συνεδρίαση, ε, εκλέγοντας στην θέση του Προέδρου, της Προέδρου μάλλον του Κοινοβουλίου του γυναίκα. Τώρα έχουμε μεγάλο αριθμό γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 288 περίπου, ε, αν και θα επιθυμούσε πολύ περισσότερες γυναίκες βουλευτές, καθώς γνωρίζουμε πόσο δραστηριοποιούνται οι γυναίκες και στην κοινωνία και στην πολιτική. Η τωρινή λοιπόν συμμετοχή των γυναικών ε, στην ε, πολιτική θα πρέπει και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε εθνικό και πάνω απ' όλα σε ευρωπαϊκό για μας να αναπτυχθεί περισσότερο γιατί προς το παρόν είναι ανεπαρκής. Πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα ψηφίσματά του έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διάφορες βάσεις, διαφορετικές βάσεις, εμπειρίες, παραδόσεις με τις οποίες μπορούν οι γυναίκες να συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων, την διατύπωση νέα θεματολογία στην πολιτική ημερήσια διάταξη των κοινωνιών μα και στην νέα αντιμετώπιση των γενικών ή παλαιότερων πολιτικών ζητημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψη αποφάσεων αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο για την, ε, αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην ε, ανάπτυξη και εξέλιξη των κοινωνιών μα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει στην διαδικασία λήψη αποφάσεων μέσα στην πολιτική, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό, όπω και σε διεθνέ επίπεδο, να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών και να υποστηριχθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλέ φορέ υπογραμμίσει τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν εν τα πολιτικά κόμματα, τα οποία καλούνται να ε, παραμερίσουν τα όποια εμπάωδια βρίσκονται στην ε, πρόοδο, στην ιεραρχία των ε, γυναικών και την εξασφάλιση βέβαια και να εξασφαλίσουν ε, με τον τρόπο αυτό ισότιμη μεταχείριση και στις ευκαιρίες για άντρες και γυναίκες. Το Δεκέμβριο του 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επί παραδείγματα, ενέκρινε μια έκθεση για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, όπου καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν μέτρα για τη βελτίωση της Συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει σε ποσοστιαία αναλογία ε, περισσότερες τώρα γυναίκες ε, βουλευτές. Όταν η ΕΚΑΦ το 1972 είχε 6% ε, γυναίκες. Στο 1971 το 1979 με το πρώτο εκλεγμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε 29% και τώρα έχει 31% γυναίκες μέλη. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ότι λίγο πολύ υπάρχει αναλογία του 30% ένα στους τρεις δηλαδή είναι γυναίκες. Το ίδιο γίνεται και στα πολιτικά μας, στις πολιτικές μας ομάδες και στις ηγετικές τους θέσεις έχουν ε, γυναίκες ε, προέδρους ή αντιπροέδρους. Έχουμε πέντε αντιπροέδρους από, τις, από τους 14, μία κοσμήτορ η οποία μάλιστα βρίσκεται εδώ παρούσα η κυρία Λούλινγκ και 14 επικεφαλής αντιπροσωπιών. Αντιπροσωπεία σημαίνει μια ομάδα βουλευτών που ανήκει μέσα σε μια πολιτική ομάδα και που προέρχονται από συγκεκριμένο κράτος μέλος. Επίσης πολυάριθμες είναι και οι γυναίκες πρόεδροι ή αντιπρόεδροι των ε, πολιτικών ε, επιτροπών ή υποεπιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να σημειώσω ότι πέραν της Επιτροπής ε, των Δικαιωμάτων της Γυναίκας και της Συμμεταχείρισης των ε, Φύλων έχουμε και την ε, Επιτροπή των Οικονομικών, Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας και προστασίας των καταναλωτών Ιεσωτερικής αγοράς Τρει ακόμη πολύ σημαντικέ δηλαδή επιτροπέ, των οποίων ηγούνται γυναίκε, βρίσκονται στην θέση του Προέδρου γυναίκε. Οι γυναίκε λοιπόν δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά στην πολιτική σε τομέα που, ή σε τομείς συγκεκριμένα που παλαιότερα ήταν αποκλειστικότητα των ανδρών. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η σε συγκεκριμενα που παλαιοτερα ηταν αποκλειστικοτητα των ανδρων επισης την σημαντικη ειναι η συμμετοχη των γυναικων στη διαδικασία του εκλέγην από το 1979 και ε, επέκεινα να ε, ε, εξελιχθεί, να αναπτυχθεί, γιατί είναι χαμηλότερη η προσέλευση των γυναικών στην κάλπη και ελπίζουμε ότι μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε με θετικά μέτρα, με ενθάρρυνση των γυναικών να προσέλθουν στην ε, κάλπη το φαινόμενο αυτό να ανατραπεί, έτσι ώστε να έχουμε ισότιμη και συμμετοχή ή άσκηση του δικαιώματος του εκλέγινα Κυρίε και κύριοι, πριν από 100 χρόνια, 15.000 γυναίκες κατέβηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, διεκδικώντας δικαιώματα και αναγνώριση των δικαιωμάτων τους. Έκτοτε η αναγνώριση και προσοχή των δικαιωμάτων των γυναικών, όπω και η προαγωγή τη ισότιμης της και των ισών δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, έχουν προχωρήσει πολύ. Πολλά όμω ακόμη μένουν να γίνουν για να εξασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των φύλων, που αποτελεί και πρέπει να αποτελεί πάντοτε ένα καθήκον βασικό που θα εγγράφεται σε κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε διεκδικεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την σημερινή διάσκεψη όπου συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες από τα Εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε πιστεύω να αποδείξουμε ότι η γυναίκα έχει τον ρόλο που της αξίζει και πρέπει να διεκδικεί τον ρόλο αυτό τόσο ως ψηφοφόρος όσο και ως πολιτικός. Ασκούσα το δικαίωμα του εκλέγην ή του εκλέγεστε. Με τη χαρά αυτή λοιπόν που έχω να βρίσκομαι μαζί σας, κηρύσω την των εργασιών σας, σας εύχομαι καλή επιτυχία και πολύ καλές και επικοδομητικές συζητήσεις. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Eh, eh, Πρόεδρε, αγαπητέ Hans Γκέρτ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και για την επίσκεψή σου εδώ στη σημερινή μας συνεδρίαση στη διάσκεψη αυτή για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας η παρουσία σου ιδιαίτερα προσδίδει κύρος στην διάσκεψή μας. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ επίσης για το μήνυμα που αποστέλεις με την ε, παρέμβασή σου και θα ήθελα να επισημάνω ότι είχαμε προσκαλέσει αρκετές ομάδες βουλευτών από τα εθνικά ε, κοινοβούλια. Ε, ιδιαίτερος λοιπόν με την παρουσία όλων εδώ των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει σημασία το μήνυμα που απέστειλε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι προάγουμε το ρόλο της γυναίκας και πάνω απ' όλα την ε, επιδίωξη της ισότιμης με συμμετοχή των γυναικών και στις ευρωεκλογές. Για εσάς, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ε, το όλο πλέγμα των σχέσεων και των πολιτικών που μπορείτε να παρακολουθείτε από τη θέση αυτή τον περίπλοκο ενδεχομένω συσχετισμών μέσα στην κοινωνία και την πολιτική. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για τα λόγια σας. Και τώρα επιτρέψτε μου και εγώ από πλευράς μου να σας καλωσορίσω. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών θεωρεί ε, άκρο σημαντική την σημερινή διάσκεψη και το θέμα της, το οποίο βέβαια πάντοτε είναι επικαιρότητα. Εφέτος λοιπόν η ε, επιλογή του θέματος ασφαλώς στηρίχθηκε στην προοπτική των ευρωεκλογών. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πέτερινγκ λοιπόν για την παρουσία του. Θα πρέπει να χαιρετήσω και να καλωσορίσω επίσης εδώ και την κυρία Βάλστρομ, τον κύριο Σπίτλα, τους επιτρόπους και τους ε, όλους τους εκπροσώπους εδώ των ε, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάσκεψη τη σημερινή βέβαια δεν συμμετέχουν μόνο πολιτικοί. Έχουμε και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε την κυρία ε, πρόεδρο της ε, οργάνωσης για τα δικαιώματα, της Εθνούς Οργάνωσης για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Έχουμε την Τουρκία καλά Υπουργό για τα δικαιώματα των γυναικών και τα θέματα της ε, οικογένειας και πολλούς άλλους εκπροσώπους. Πολλά θέματα λοιπόν που θα μας προσφέρουν σήμερα θα έχουν να κάνουν και με, την, ε, και με τις ίσες ευκαιρίες και με τις ε, δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν αυτές οι προσεχείς ευρωεκλογές. Περιμένουμε ακόμα τον κύριο Κούρσα ο οποίος ε, όπου να είναι θα έρθει, από ό,τι ενημερώνομαι. Και ω εκ τούτου θα παρακαλέσω την κυρία Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, που είναι επιφορτισμένη και με τις διοργανικές σχέσεις και με την στρατηγική ε, της επικοινωνίας, την κυρία Βάλστρομ, να μας πει δύο λόγια. Ο Σπίτλα ασχολείται με τα θέματα της ε, απασχόλησης, ε, τα εργασιακά και βέβαια την συμμεταχείριση ε, ανδρών και γυναικών, την ισότητα ευκαιριών. Επίσης θα ακούσουμε συναδέλφους, κυρίως γυναίκες, που θα μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καλώς ορίζω εδώ την κυρία Αστριτ την παλαιότερη εν ενεργεία ευρωβουλευτή, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 1965, και πιστεύω ότι θα έχει πολλά να μας πει από τις εμπειρίες της. Επίσης η κυρία Ζήτα η οποία εκπροσωπεί το διοργανικό δίκτυο βουλευτών, ένα άτυπο δίκτυο μεν, πολύ σημαντικό όμως για την ε, εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Κατά τη διάρκεια της ε, διάσκεψής μας θα ακουστεί και μια μελέτη που θα παρουσιαστεί, μια μελέτη την οποία έχει παραγγείλει η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών, και που αφορά τις ποσοστώσεις στην εκλογική διαδικασία υπέρ των γυναικών ανάλογα με το πώς εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος. Η κυρία Ντάλερουπ, η κυρία Ντρούντε Ντάλερουπ από το Πανεπιστήμιο του Στοκχόλμης θα μας κάνει τη σχετική παρουσίαση. Και βεβαίω, κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, περιμένουμε να ακούσουμε και τι δικέ σα εμπειρίε και απόψει για τα όσα έχετε δει και στι πατρίδε σα και στα δικά σα κοινοβούλια. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσία εδώ και επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην ε, κυρία Επίτροπο, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Μαρκότ Βάλστρομ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι χαρούμενη και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να γιορτάσουμε τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας. Ακούσατε από τον Πρόεδρο Πέτερη ότι είναι μια εξαιρετική χρονιά για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία με τις ευρωεκλογές ε, τον Ιούνιο. Στην Ευρώπη το 52% του πληθυσμού είναι γυναίκες. Για μένα λοιπόν φαντάζομαι και για πολλούς από εσά το να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται ισότιμα στις συζητήσεις, ε, στις αποφάσεις, ε, είναι θέμα καθαρά δημοκρατίας. Θα ήθελα πολύ σύντομα να μιλήσω για τρία θέματα. Καταρχάς τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στην Ευρώπη σήμερα. Η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τι κάνουν για τις γυναίκες και οι γυναίκες τι μπορούν να κάνουν για τον εαυτό τους και για την Ευρώπη. Θα ήθελα με λίγα παραδείγματα να προσπαθήσω να σας ε, δείξω τι μπορεί να σημαίνει σήμερα το να είσαι Ευρωπαία γυναίκα. Ας ε, ξεκινήσουμε με την 22χρονη Ορτινέτα, η οποία είναι φοιτήτρια μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Ρήγας. Το μεγαλύτερο δίλημά της είναι το αν θα δεχτεί μία προσφορά από μια εταιρεία λετωνική α, στη Λετωνία ε, στον τομέα των υπολογιστών για να θα τελειώσει το μάστερ της. Προς το παρόν, ε, αποκλείεται να της δώσουν τόσα λεφτά όσα στο φίλο της. Οι γυναίκες σήμερα πληρώνονται κατά 16% λιγότερο από τους άντρες για την ίδια ακριβώς δουλειά με τους άντρες. Στην Εστονία αυτό το χάσμα είναι πάνω από 22% η διαφορά των μισθών μεταξύ των ανδρών και γυναικών ε, στην Ευρώπη κλείνει σιγά σιγά, αλλά θα χρειαστούν περίπου 100 χρόνια ακόμα για να πληρώνονται οι γυναίκες το ίδιο με τους άντρες για την ίδια δουλειά. Κι όμως, ο ίσος μισθός για ίδια εργασία είναι ένα δικαίωμα το οποίο εγγράφεται στις ευρωπαϊκές ε, συνθήκες. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Το 2006 η Λόνα, που είναι μια ε, Ουγγαρέζα από την 26 χρονών, ζήτησε μία δουλειά σε μία μικρή εταιρεία. Προσλήπη της, της είπαν ότι δεν είναι επιλέξιμη γιατί μόνο άνδρες θα μπορούσαν να προσληφθούν σε αυτή την εταιρεία. Της πρόσφεραν μια δουλειά καθαρίστριας που θα της απέφερε πολύ λιγότερα. Η αρχή για την ίση μεταχείριση της Ουγγαρίας ε, αποφάσισε υπέρ της Ιλώνας και η εταιρεία πλήρωσε ένα μικρό πρόστιμο. Η Ιλώνα όμως δεν θα πάρει καμία αποζημίωση. Αλλά όταν ε, ε, ξεκίνησε να λειτουργεί η, εταιρεία αυτή και, και με άλλα υποκαταστήματα, ε, της πρόσφεραν μία, τη δουλειά που είχε ζητήσει. Επίσης, σε μία εταιρεία consultancy, μία άλλη γυναίκα στη Γερμανία, ε, είχε παιδιά Είχε πρόβλημα όμως με τα παιδιά της, δεν έβρισκε κάποιον να τα φροντίσει και επομένως σταμάτησε να δουλεύει ε, γιατί δεν μπορούσε να βρει κάποιον να τα φυλάει. Φανταζόμασταν ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες ε, αποζημιώνουν και τιμούς, τιμούν τις γυναίκες που κάνουν παιδιά καθώς ε, οι πληθυσμοί μας γυράσκουν. Αλλά στην πραγματικότητα ακόμα και πλούσιες χώρες όπως η Γερμανία δεν έχουν δικαιώματα δεν είχαν δικαιώματα ε, για την άδεια μέχρι να τους υποχρεώσει η Ευρώπη να το κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες ε, δύσκολα τα καταφέρνουν με ταχυδακτηλουργικό τρόπο μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και της οικογενειακής ζωής. Συχνά η γέννηση των παιδιών ε, συνιστά μειονέκτημα, πρόσκομα ε, για αυτές όταν θέλουν να ζητήσουν ε, θέση στην αγορά εργασίας. Επίσης αυτές οι γυναίκες που σας ανέφερα όταν πάρουν σύνταξη θα έχουν ε, χαμηλότερη σύνταξη από τους άντρες. Επίσης μία από τις τρεις γυναίκες ε, λένε οι στατιστικές ότι θα έχουν προβλήματα φυσικής βίας ή σεξουαλικά προβλήματα ε, στο χώρο εργασία τους. Επομένως, όπως είπε και η Σιμόντε Μποβουάρ, εξακολουθούμε να ζούμε σε έναν κόσμο ανδρών. Τώρα, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες για αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πραγματικά κάνει πολλά πράγματα για τις γυναίκες. Απαγορεύεται η διάκριση εις βάρος των γυναικών και στις συνθήκες και στη Χάρτα ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Από την δεκαετία του 70 οι ευρωπαϊκοί νόμοι έχουν ε, επεκτείνει τις ε, επιλογές των γυναικών και βελτίωσαν τη ζωή τους. Το ποσοστό των γυναικών στην δουλειά έχει αυξηθεί. Είναι περίπου τώρα το 59% επίσης των αποφύτων στα πανεπιστήμια. Η Κομισιόν έχει νομοθεσία για να ενδυναμώσει το δικαίωμα στην άδεια μητρότητας και έχουμε συστήσει δράση για να υπάρχουν περισσότερες εγκαταστάσεις για τη φύλαξη των παιδιών. Οι κοινωνικοί εταίροι, και φαντάζομαι ότι ο Βλαντιμίρ θα μιλήσει περισσότερο για αυτό το θέμα, ε, θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθεί η σχετική οδηγία και θα ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο το Μάιο για την, την ισότητα. Επίσης, το Ινστιτούτο για την Ίση Μεταχείριση θα συνεισφέρει στην αφύπνιση του κοινού ε, για τα θέματα ίσης μεταχείρισης. Το πρόγραμμα Δάφνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βοηθάει τους ε, τοπικούς φορείς και τις τοπικές αρχές να καταπολεμήσουν την βία στο σπίτι και να προστατεύσουν τα θέματα. Έχουμε καλές νομοθετικές αρχές νομοθετικά κείμενα, αλλά αυτό δεν αρκεί. μπορούμε να επεκτείνουμε την νομοθεσία μας Πάντως, οι απόψεις των γυναικών μπορούμε να πούμε ότι λαμβάνονται υπόψη. Το τρίτο ερώτημα. Τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες τώρα για τον εαυτό τους και για την Ευρώπη. Οι γυναίκες στην Ευρώπη επί δεκαετίες είχαν το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Αλλά θα πρέπει να πολεμήσουμε, χρειάστηκε να πολεμήσουμε πολύ για αυτά τα δικαιώματα. Η πρώτη χώρα που κερδίθηκε αυτή η νίκη ε, πριν από πάνω από 100 χρόνια ήταν η Φιλανδία, που έδωσε αυτά τα δικαιώματα σε όλες τις γυναίκες, ανεξάρτητα από την τάξη του, τη φυλή τους κτλ. Ε, σε άλλε χώρε όμω χρειάστηκαν περισσότεροι αγώνες και περισσότερα χρόνια. Βέβαια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα στι ε, κυβερνήσει και στα ε, κοινοβούλια των 27 ε, κρατών μέλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το λιγότερο το 1 τέταρτο των υπουργών είναι γυναίκε και των βουλευτών. Τώρα, τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι φέτος η 300 η επέτειος από την πρώτη ε, καθολική εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όμως μόνο το 1 τρίτο ε, σήμερα είναι, γυναίκες, είναι βουλευτίνες. Επίσης ποτέ δεν υπήρξε ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γυναίκα. Σήμερα ε, η Κομισιόν έχει πολλές γυναίκες, ε, αλλά όμως δεν είναι πάνω από 10, 10 στις 27. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το μισό του πληθυσμού ε, υποεκπροσωπείται. Δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι καλοί άνθρωποι, παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Ε, δεν είμαι θεροβάμων. Αλλά αν οι γυναίκες εκπροσωπούνται ισότιμα εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ε, τότε θα λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα θέματά του, Δεν θα προωθούν οι άντρε τα δικά του θέματα. Οι γυναίκε έχουν εμπειρία, έχουν γνώσει κτλ. Τα προβλήματα που έχουν ε, υποστεί οι γυναίκε που σα ανέφερα θα αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερο ζήλο ε, και συντομότερα αν υπήρχε ίσως αριθμός ανθρώπων και γυναικών ε, στα όργανα λήψη των αποφάσεων στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Η τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης επίσης θα πρέπει να έχουν περισσότερες γυναίκες υποψηφίους ε, στις εκλογές. Ιδανικά θα ήθελα να υπάρχει ίσως ε, αριθμός ανδρών και γυναικών σε κάθε κόμμα, σε κάθε κοινοτική χώρα. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα ε, σε ό,τι αφορά τους πολιτιστικούς και νομικούς όρους. Αλλά είτε η νομοθεσία δεν προβλέπει ποσοστώσεις, είτε δεν υπάρχει αρκετή πίεση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει πίεση από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει έλλειψη καλών ε, γυναικών υποψηφίων. Η πραγματικότητα από την ιστορική εμπειρία ε, δείχνει ότι οι άντρες τείνουν να διαλέγουν τους άντρες. Επίσης θα θέλαμε να θαρρύνουμε τις γυναίκες να ψηφίσουν και να υπάρχει πιο ε, ισομερής ε, εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε η δημοκρατία να είναι 50% άνδρες, 50% γυναίκες. Ε, η Μέρι Ρόμπινσον, η Βιβιάννα Ιντόλ, πολλές ε, γυναίκες ε, επίτροποι και πολλές άλλες γυναίκες είναι υπέρ αυτής της ιδέας. 50% άνδρες, 50% γυναίκες. Ε, επομένως, αγαπητές ε, φίλες, Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν απόκειται μόνο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν την ισότητα. Υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, και πολλών οργανώσεων γυναίκες. Καθένας από εμά εδώ σήμερα θα πρέπει να ενθαρρύνει τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τις ψήφους τους και να ορθώσουν το ανάστημά τους για να υπάρξει ίση εκπροσώπηση ε, στο επόμενο κοινοβούλιο, στην επόμενη επιτροπή και εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ελπίζουμε με τη νέα συνθήκη όταν επικυρωθεί να βοηθήσει και αυτή προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο καθένας από εμά μπορεί να εξηγήσει ότι οι γυναίκε των γυναικών θα πρέπει επίσης να μετρήσουν στην Ευρώπη, όπως και των ανδρών. Σήμερα η Κομισιόν ε, ξεκινάει μία συζήτηση για τις γυναίκες της εκλογέ στην ιστοσελίδα μας για τις εκλογέ. Ε, αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι τις 25 Μαρτίου και ελπίζω πολλές από εσά ε, να συμμετάσχετε και να φέρετε αυτή τη συζήτηση στους ε, δρόμους ε, και στις πλατείες της Ευρώπης. Φυσικά σήμερα εστιάζουμε στην Ευρώπη, αλλά τα δικαιώματα των γυναικών διακυβεύονται παντού. Στις 7 και 8 Μαρτίου θα συμμετάσχω στο Διεθνές Συμπόσιο για την ηγετική θέση των γυναικών για την ασφάλεια και την ε, ειρήνη που οργανώνεται στη Μονρόβια από την Λιβερία και από τον ε, Τάρι Χάλανεν, πρόεδρο της Φιλανδίας. Μία γυναίκα είπε ότι πάνω από το 50% του, του παγκόσμιου πληθυσμού είναι γυναίκες. Κι όμως, επί πολύ καιρό, ε, τα ενδιαφέροντα των γυναικών, τα συμφέροντα των γυναικών, οι ανάγκες των γυναικών, η φωνή των γυναικών δεν έχουν ακουστεί δεν αποφασίζουν ποιο θα μα κυβερνήσει. Δεν καθοδηγούν αυτού που κυβερνούν. Μια και οι γυναίκες είναι από του πιο αδύναμους πολίτες, με λιγότερες οικονομικές ε, δυνατότητες και κοινωνικούς πόρους, θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, ούτως ώστε να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή τους. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δράσουμε. Αυτές οι εκλογές ας γίνουν μια πραγματική ευκαιρία για να προωθήσουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο στις Ευρωπαϊκές Δημοκρατίες. Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Σπίτλα. Βλάντιμιρ Σπίτλα, Επίτροπο για θέματα απασχόλησης, κοινωνικές υποθέσεις και ίσες ευκαιρίες. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι που είμαι εδώ ανάμεσά σας για την ε, Παγκοσμίου ημέρα της γυναίκας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που με καλέσατε για τη συνάντηση αυτή. Να σας πω θα επιθυμούσα ότι είναι για μένα μία τιμή πραγματική Έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για αυτήν την τιμή. Χάρη στο διάλογο αυτό μπορούμε να συνεργαστούν τα μεμονωμένα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συζήτηση αυτή να αποβεί σε κάτι το πραγματικά αποτελεσματικό. Η ισότητα μεταξύ άνδρων και είναι βασική αξία Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Οι ανεπτυγμένε κοινωνίε οικοδομήθηκαν ακριβώ βάσει της ισοτιμίας αυτών, αυτής μεταξύ όλων των πολιτών της. Και είναι μια αυτή καθ' αυτή αξία, όχι για ορισμένες χρήσεις και επιδιώξει. Και είναι κάτι το θετικό να έχουμε αυτή την ε, ισοτιμία ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες. Έστω και αν δεν είναι πραγματική αυτή η ισότητα, εμείς πάντως θα δώσουμε τη μάχη μας για να την πετύχουμε. Πρόκειται και η αξία και η ηθική, αλλά και όσον αφορά τις επιδιώξεις μας. Αυτή η βασική αξία στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή οφείλεται στην υποστήριξη πάνω απ' όλα των κυβερνήσεων των κρατών μελών, όπως επίσης και των βουλευτών τους. Έχουν σημειωθεί πρόοδοι στον τομέα αυτό και εμείς καταβάλαμε προσπάθεια ώστε κάθε πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσέχει και το θέμα της εκπροσώπησης των γυναικών και των ανδρών βέβαια. Στις κοινωτικές πολιτικές αυτό το στοιχείο για το φύλλο είναι κάτι το βασικό σε κοινωτικό επίπεδο επαναλαμβάνουμε. Κανείς δεν μπορεί να νιωθεί το γεγονός ότι η εκπροσώπηση των γυναικών είναι αρκετά πιο ισορροπημένη από ό,τι στο παρελθόν. Θα μπορούσα να σας αναφέρω αρκετά παραδείγματα αρκετά περισσότερες γυναίκες που απασχολούνται και έχουμε πάνω από το 56%, 60% πια που αναφέρεται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια χρειάζεται ένας έλεγχος γιατί η σημερινή οικονομική κρίση θα μπορούσε να ε, χειροτερεύσει δυστυχώς την κατάσταση της απασχόλησης γυναικών. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα προσπαθήσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι γυναίκες να εκπροσωπούνται πραγματικά και να υπάρξει μια κατάλληλη αντιμετώπιση της κρίσης. Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευση των γυναικών είναι πολύ ανώτερο, πολύ ψηλότερο από ό,τι στο παρελθόν το 60% των πολιτών της Ευρωπαϊκής με πανεπιστημιακά διπλώματα είναι γυναίκε. Άρα λοιπόν έχει επιτευχθεί πρόοδος, αλλά σε διάφορους τομείς επίσης οι γυναίκες δυστυχώς μειονεκτούν απέναντι στους άνδρες. Διαφορά αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. 17 περίπου της 100 αυτή η διαφορά υπέρ των ανδρών. Τι 3 Μαρτίου γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα μια νέα εκστρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος αυτού του προβλήματος και υπολογίζω στην συνεργασία σας, την προσπάθειά σας για να μπορέσουμε και εκεί να σημειώσουμε βήματα προς τα εμπρός και πρόσβαση γυναικών σε θέσεις υπεύθυνες, υψηλές. Ε, αυτό είναι και το σημερινό μας θέμα. Άλλωστε, η παρουσία στα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών, η παρουσία των γυναικών είναι περίπου 24% και στις κυβερνήσεις επίσης δεν ε, υπάρχει κάτι καλύτερο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι γυναίκες εκπροσωπούνται με ένα ποστό του 31% κάπως υψηλότερο, αλλά από το 1999 δεν έχουμε μια βελτίωση αυτού του ποσοστού. Οι εκλογές λοιπόν του 2009 αποτελούν μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ελπίζω δε ότι δεν θα αφήσουμε να ξεβγεί από τα χέρια μας η ευκαιρία αυτή. Για να δούμε τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιριών είναι μόνο περίπου στο 11%. Κατά την άποψή μου δεν πρόκειται για μια κακή διαχείριση και χάνεται ποσοστό εξυπνάδας ακριβώς ε, των γυναικών. Και τα αποτελέσματα σε αυτό το τομέα μπορούμε να σας πούμε ότι είναι περιορισμένα. Χάρη όμως πάνω χάρη στο παράδειγμα της Νορβηγίας. Εκεί πάνω από το 40% των γυναικών είναι στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών. Είναι 40% επαναλαμβάνω γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και βλέπουμε έτσι ότι μπορεί τάχιστα να αλλάξει η κατάσταση χάρη σε ρυθμίσεις και νομικής φύσεως υπέρ της αντιμετώπιση αντιμετώπισης των δύο φύλων να υπενθυμίσουμε ότι από τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία στα πλαίσια της προσπάθειάς μας ε, για ίσες ευκαιρίες για τα δύο φύλλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε Έκανε γνωστή μάλλον μια νέα έκθεση εμπειρογνωμόνων, είναι στη διάθεσή μας, που κάνει μια ανάλυση των γυναικών στα πλαίσια της πολιτικής αλλά και σε άλλους τομείς. Τι αποδεικνύει αυτή η έκθεση ότι στις θέσεις κλειδιά της πολιτικής ε, υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες και τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να καταβάλουν ακόμα περισσότερες προσπάθειες ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και η κατανομή της εξουσίας ε, θα πρέπει να αλλάξει αυτή επίσης εκτός από την πολιτικό τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Πεπισμένος είμαι ότι χρειάζεται να προσπαθήσουμε ιδιαίτερα για να πετύχουμε να προσφέρουμε σε ευκαιρίε και στα δύο φύλλα. Μια περισσότερο ισορροπημένη εκπροσώπηση άνδρων και γυναικών σε υπεύθυνε θέσει είναι μια προπόθεση για μια συντοποιημένη δημοκρατία, αποτελεσματική δημοκρατία και η νευμάρια τη οικονομία μα. Όλο και περισσότερο μελέτε τι αποδεικνύουν ότι η σχέση είναι θετική από την εκπροσώπηση των γυναικών σε μια εταιρεία, σε μια επιχείρηση και στο ποσοστό επιτυχίας της εταιρεία αυτής. Δεν είναι ικανοποιητικό λοιπόν το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε αυτές τις θέσεις λήψης αποφάσεων και πέρυσι δημιουργήθηκε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ε, συγκεντρώνει τα σημερινά ευρωπαϊκά δίκτυα που έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό και ο στόχος ποιος είναι να συνειδητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο στην κοινή γνώμη τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα. Το 2009 αποτελεί σημαντική χρονιά και λόγω των ευρωεκλογών αλλά και για τις γυναίκες. Οι εκλογέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι σημαντικές θέσεις, ποιος θα τις καταλάβει, για τα κράτη-μέλη, για όλους εκείνους οι οποίοι ε, συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες που προτείνουν, ορίζουν ή εκλέγουν, έχουν αυτή την ευθύνη ότι θα πρέπει να επιλεχθούν και γυναίκες για αυτές τις θέσεις. Υπάρχουν αρκετές υποψήφιες γυναίκες, αλλά τα συστήματά μας δεν τους προσφέρουν την κατάλληλα ευκαιρία, δεν τους ανοίγουν το δρόμο για να πετύχουν τις φιλοδοξίες τους ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Στα ψηφοδέλτια χρειάζεται να συμμετάσχουν και πολλές γυναίκες. Ε, εντάξει υπάρχουν αρκετές αλλά δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει να είναι σε εκλέξιμε θέσει ε, τα ονόματά του, υποψηφιότητέ του, για να καταλάβουν αυτέ τι υπεύθυνε θέσει. Και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ελέγξουν το δικό του το εκλογικό σύστημα που να μην παρεμποδίζει τι γυναίκε, να μην του κλείνει το δρόμο τη πολιτική και να θετήσουν τι κατάλληλε πολιτικέ ρυθμίσει ε, όπω με την ε, θέσπιση νόμων που να μην ευνοούν την υποεκπροσώπηση γυναικών στην πολιτική και στα ψηφοδέλτια των ε, πολιτικών κομμάτων χρειάζονται περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν από ό,τι στο παρελθόν. Επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι να επιβεβαιώσω ακόμα μια φορά την προσπάθεια και της Επιτροπής και τη δική μου την προσπάθεια ε, για μια προσφορά ίσων ευκαιριών στα δύο φύλλα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, όπως ακριβώς προβλέπεται και από το πρόγραμμά μας για την δημιουργία αυτών των ίσων ευκαιριών. Ελπίζω ότι την ευκαιρία αυτή δεν θα τη χάσουμε από τα χέρια μας για το 2009 που θα μπορούσε να πετύχει μια βελτίωση καταστάσεως και μια ισορροπία στην εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε υψηλές υπεύθυνε θέσεις σημαντικό ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια όπως επίσης και το Ευρωκοινοβούλιο και θα ήθελα μαζί να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και θα ήθελα εδώ να ε, καλωσορίσω τον εκπρόσωπο της Τσεχικής Δημοκρατίας, τον κύριο Υπουργό για Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εθνικές Μειονότητες, Μιχαήλ Κότσαπ. Του δίνω το λόγο λοιπόν, ευθύς αμέσως. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. <clears throat> Takže vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, Πρόεδρε. κύριε επιτρόπε, κύριε επιτρόπε, κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου εδώ να εκφράσω την απόψή μου και μάλιστα σύντομα σχετικά με τα θέματα αυτά που είναι ιδιαίτερα επίκαιρα. Λόγω και των προσεχών ευρωεκλογών. Ίσως ορισμένα πράγματα που υπήθηκαν από τον Επίτροπο Σπίτλο θα τα επαναλάβω και εγώ. Αλλά ξεχωριστά προετοιμάσαμε τις εισηγήσεις μας, γι' αυτό ίσως συμπίπτουμε σε περικά σημεία και αυτό που δείχνει άλλωστε ότι έχουμε κοινέ απόψεις σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, Διεθνή ημέρα γυναικών. Ξέρετε ότι ξεκινήσαμε από τη σκέψη να πρώτα απ' όλα να έχουν ε, δικαίωμα ψήφου γυναίκες και ήταν, ε, ήταν δύσκολος ο δρόμος. Οι γυναίκες πραγματικά κατέκτησαν το δικαίωμα αυτό. Τι γίνεται όμως τον, το θέμα του εκλέγεστε. Εδώ παρόλο που υπάρχουν ρυθμίσεις ε, νομικές πολιτικές, ε, από την πολιτικής πλευράς αυτός είναι ένας τομέας σχεδόν καθαρά ανδρικός. Οι άνδρες καθορίζουν τις πολιτικές προτεραιότητες και η πολιτική προσανατολίζεται στους άνδρες Υπάρχουν αρκετά εμπόδια που παρεμποδίζουν ακριβώς τις γυναίκες να φτάσουν σε υψηλές θέσεις λήψης αποφάσεως πολιτικές κλπ. Από τα κύρια εμπόδια είναι ότι υπάρχουν αντιλήψεις αρνητικές βάσει των οποίων οι γυναίκες θα πρέπει μάλλον να παραμένει με τα παιδιά της, στην κουζίνα της, να δημιουργεί τις βάσεις για ε, την οικογένειά της και θα πρέπει ο άνδρας να κερδίζει τα νέα και από θεσμικής πλευράς ε, έχουμε το σύστημα πρόσβασης στις εκλογές και την επιλογή ανδρών και γυναικών στα πολιτικά κόμματα. Εδώ οι εκλογές κυρίως διεξάγονται βάσει συμμετεχόντων, βάσει υποψηφιότητων στο ψηφοδέλτιο και οι πολίτες από την ξεκίνημα ήδη έχουν μια περιορισμένη δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να δούμε αυτό το σύστημα επιλογής υποψηφίων στο ψηφοδελτίο. Και αυτό είναι το, αυτός είναι ο κύριος τομέας τον οποίο θα πρέπει να επιδράσουμε, να επηρεάσουμε για την συμπερίληψη γυναικών. Ε, από την μια μεριά έχουμε κάποιες, αρκετές μάλλον υποψηφιότητες, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουμε συμμετοχή γυναικών στις κυβερνήσεις. Ο Επίτροπος Πίδλα μίλησε για το 30% των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 37% στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν Επίτροπη. Γυναίκες και στα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το 24% γυναίκες εκλεγμένα μέλη. Υπάρχει μια ίση εκπροσώπηση αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ίση εκλογή. Ε, αρκετές γυναίκες ε, καταβάλουν προσπάθειες ε, για τις ίσες αυτές ευκαιρίες σε και γυναίκες ε, και με διάφορες ενέργειες έχουν δραστηριοποιηθεί Έχουμε την πλατφόρμα του Πεκίνου και την επέλευση των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται για την πολιτική παρά την άποψη πολλών σχετικά με το αντίθετο και υπάρχουν ε, αποδείξεις ε, αυτών ε, και γυναίκες σε κοινοτικό επίπεδο, δημοτικά συμβούλια κλπ. Συμμετέχουν αρκετές γυναίκες. Οι γυναίκες σε υψηλές υπεύθυνες θέσεις πολιτικής, κυρίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σιγά σιγά η θέση τους βελτιώνεται. Σιγά σιγά όμως. και είναι η ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για τα ψηφοδέλτια, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμα φορά, για να μπορέσουμε να παρακάψουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ε, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά στην πολιτική. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια εξήμιση της καταστάσεως από εντελώς διαφορετική οπτική γωνία. Οι γυναίκες πρέπει να συμμετάσχουν στην ε, προετοιμασία για την πολιτική ζωή και τα πολιτικά κόμματα όμως τελικά αποφασίζουν ποια θα είναι αυτά τα ψηφοδέλτια, ποιοι θα συμμετάσχουν, ποιοι θα συμπεριληφθούν σε αυτά τα ψηφοδέλτια, ποιος θα έχει δυνατότητα να εκλεγεί ή όχι. Και το θέμα των ποσοστώσεων ε, στα ψηφοδέλτια γυναικών, τη συμμετοχή τους αυτή. Εκεί ασκείται αρκετές φορές μια κάποια κριτική. Παρόλε τις ε, προσπάθειες αρκετές ή ε, τουλάχιστον για δέκα χρόνια θα υποεπροσωπούνται οι γυναίκες στην πολιτική ζωή οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πολλοί άλλοι φορεί θα πρέπει να καταλάβουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προωθήσουν ε, τη συμμετοχή γυναικών και πρόκειται για μια μακρόπνοη προσπάθεια και πολιτική και θα πρέπει να ξεπεραστούν ε, οι παλιές αντιλήψεις περί του θέματος και στα κράτη όπου συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες ε, στην πολιτική, οι χώρες αυτές έχουν πετύχει το στόχο τους μετά από μια μακρά σειρά ετών συνεργασίες ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στα κοινοβούλια και στη συμμετοχή γυναικών, τη συμπερίληψη γυναικών στα ψηφοδέλτια όπως είπαμε. Και ακόμη Εδώ το πρόβλημα είναι πώς θα προσφέρουμε κίνητρα στις ε, πολιτικές ομάδες, στα πολιτικά κόμματα για μια παρόμοια νέα προσέγγιση. Οι εκλογέ άνδρες και γυναίκες από τη στιγμή που επιθυμούν περισσότερη ψηλότερη προσώπηση γυναικών στην πολιτική θα πρέπει αντίστοιχα και τα πολιτικά κόμματα να αντιδράσουν, να εγκαταλείψουν πεπαλαιωμένες θέσεις, κλασικές, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις γυναίκες της 2 Μαρτίου του 2000. Υποστηρίχθηκε εκεί ε, χρήση ποσοστώσεων για να παρακάμψουμε εμπόδια που εμποδίζουν ακριβώς την συμμετοχή γυναικών όπως και των ανδρών και έχουμε ένα κατόφυλλο της τάξης του 40% σε κάθε παρόμοιο πλαίσιο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι το κατόφλι αυτό του 40% θα πρέπει να γίνει σεβαστό και στις ε, προσεχείς εκλογές, στις ευρωεκλογές. Θα ήθελα δε να καταλήξω ευχαριστώντας όλους σας, ευχαριστώντας και όλες τις γυναίκες για την καθημερινή τους δραστηριότητα και σας ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. και θα ήθελα και να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκριμένους μας από τα ευρωπαϊκά όργανα. Στο δεύτερο λοιπόν μέρος της διάσκεψης θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσά, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων ή των οργανώσεων που εκπροσωπείτε εδώ. Σε όλους εσάς που δέχτηκαν ε, την πρόσκληση και ήρθατε εδώ. Θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε γενικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα σας παρακαλέσουμε σε τούτου να περιοριστείτε στις παρεμβάσεις στα δύο λεπτά. Θα δείτε ότι έχουμε και χρονόμετρο που χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε το χρόνο και να μην επεκτηνόμαστε περισσότερο από ό,τι χρειάζεται και έτσι να επιτρέψουμε και στους άλλους συμμετέχοντες εδώ που το επιθυμούν να μιλήσουν. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Αθηνά Κωνσταντζα από την Αθήνα να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, την Ελλάδα. Από την Ελλάδα, ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αισθάνομαι κι εγώ ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι και συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα για τις ευρωπαϊκές εκλογές γιατί αποτελούν σημαντικό γεγονός εφόσον αποτελούν μια έκφραση της βούλησης των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί διαμορφώνουν συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. Είναι εκλογές ευθύνης, πρέπει να αναδείξουν τον προβληματισμό μας γιατί όλοι θέλουμε μια Ευρώπη με συνθήκες ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών και με ποιότητα ζωής για είναι επίσης σημαντικό ότι η συνάντηση σε αυτή γίνεται με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας στις 8 Μαρτίου, διότι οι γυναίκες σήμερα εργαζόμενες με διπλούς και πολλούς πολλαπλούς ρόλους ε, βρίσκονται σε ένα αντίξωο και δύσκολο και αρνητικό κόσμο να παλεύουν για την κατοχήρωση των δικαιωμάτων. Σαν πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Ελλήνων θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία όσον αφορά την ε, συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και να πω την άποψη ότι παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται ποσόστοση κατά ένα τρίτο στη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, στις βουλευτικές εκλογές, στα εθνικά όργανα, στις επιτροπές λήψης ε, αποφάσεων στην έρευνα και στην τεχνολογία, παρά τα πέραν από την νομοθεσία το σημαντικότερο είναι να αποκτήσουν εμπιστοσύνη οι ίδιες οι γυναίκες να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη απέναντι στις γυναίκες υποψήφιες οι οποίες θα προβάλλουν τα αιτήματά μας και θα υπερασπίσουν τα δικαιώματά μας. πιστεύω ότι οι περισσότερες γυναίκες που να συμμετάσχουν στα ευρωψηφοδέλτια και σε εκλόγιμες θέσεις θα είναι σημαντικές και για την προώθηση της ισότητας αλλά και για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος αλλά και για θέματα καθημερινότητας του πολίτη. το θέμα της ισότητας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασική αρχή της δημοκρατίας. Για επόμενα ζητήματα η συνάδελφός μου επίσης από την Ελλάδα η κυρία Ράπογλου θα μπορεί να τοποθετηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καρακώστα, εάν λέμε σωστά το όνομά σας και θα ήθελα να στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Τσίμερμαν, πρόεδρο της αντιπροσωπείας του Γαλλικού Κοινοβουλίου της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή την ημερίδα που στην παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών ε, σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική στιγμή και για τη Γαλλία αλλά και για όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Γιατί? Γιατί απλούστατα πιστεύω ότι στη Γαλλία όπως και σε άλλες χώρες, χάρη στην Ευρώπη, η πολιτική που προωθούν ε, τα κράτη-μέλη, οι πολιτικές υπέρ των γυναικών, ε, χάρη στην Ευρώπη επαναλαμβάνω, τα σύνορα των δικαιωμάτων έχουν εξελιχθεί, έχουν προχωρήσει. Το 1972, το 1983, το 2001 ε, ψηφίστηκαν νόμοι ε, στη Γαλλία ε, ουσιαστικά λόγω της προσπάθειας μεταφοράς των ευρωπαϊκών ε, νομοθετικών κειμένων, ε, κανονισμών και οδηγιών. Και αυτό θα ήθελα να το υπογραμμίσω. Στη Γαλλία, μόνο χάρη στο νόμο, στη δύναμη του νόμου, καταφέρνουμε ε, να προχωρήσουμε σε πολιτικό επίπεδο παραδείγματο χάρη για, τους, για τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια, υπάρχει απόλυτη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα λοιπόν, όταν ε, οι γυναίκες και οι άντρε προσφεύγουν στις καλπε εκλέγουμε 45 με 46% γυναίκες και τις στέλνουμε στην Ευρωβουλή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σπίτλερ. Γιατί, Γιατί χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα έχουμε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος επιτρέπει και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο, να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα βήματα. Οι αντιπροσωπείες των γυναικών συγκεντρώθηκαν χθες ε, 350 άτομα για να υλοποιήσουν ε, τις πολιτικές, ε, κάποιες πολιτικές ε, και να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να είναι πολύ πιο αποφασιστικές στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και τώρα επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στην κυρία Ζακλίν πρώτη αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας του, της Γαλλικής Γερουσίας για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η αντιπροσωπεία της Γερουσίας συμμετέχει στην εκδήλωσή σας αυτή για να τονίσουμε ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το θέμα και στο μέλλον σε σχέση και με τις ευρωεκλογέ, ώστε η φωνή των γυναικών να ακουστεί στο μέλλον συνειδητοποίηση και για να ψηφιστούν γυναίκες και για την εκπροσώπηση. Αυτά θα πρέπει να τα σεβαστούμε. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια. 22% των γυναικών στη Ρουσία που έχουμε εκλεγεί το Σεπτέμβριο που μας πέρασε έγινε αυτό και είπατε ότι 30% των γυναικών ε, εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα και ο στόχος είναι να πάει και μέχρι το 40%. Θα πρέπει να το προσπαθήσουμε για μια πρόοδο πραγματικά και στις μελλοντικέ εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σίγουρα και, και όπως ε, είπε και η κυρία Ζήμερμεν θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτοί οι νόμοι στις χώρες μας. Πολύ δουλειά έχουμε μπροστά μας, πολύ να προχωρήσουμε και γι' αυτό ιδιαίτερα περήφανα θα δραστηριοποιηθούμε και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ των γυναικών και θα στεφτεί η προσπάθειά μας με μεγαλύτερη ακόμα επιτυχία στις επόμενο αυτό ραντεβού στις εκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Κωνσταντε από την Ιταλική Αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομα, σύντομα. Σίγουρα και εγώ είμαι υπέρ των όσων υπόθηκαν για τις ποσοστώσεις ε, η έποψή μου είναι ότι αντικειμενικά μιλώντας έτσι στις διάφορες χώρες όπου υιοθετήθηκαν τα μέτρα αυτά είχαμε αρκετά βήματα προς τα εμπρός και η Ευρώπη ιδιαίτερα βοήθησε όπως είπε και εκπρόσωπος του Γαλλικού Κοινοβουλίου στην όλη αυτή διαδικασία και αυτό ακόμα περισσότερο θα πρέπει να γίνει. Στα πλαίσια αυτής της οικονομικής κρίσης που περνάει η Ευρώπη φοβάμαι ότι ε, όλα αυτά θα πάνε εις βάρος των γυναικών, πολλά τουλάχιστον από αυτά. Και το θέμα και της εκπροσώπησης. Ε, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της κοινωνικής και της οικονομικής κρίσης ε, και αυτό θα μπορούσε να επανέλθει με μια πιστοδρόμηση ιδιαίτερη τουλάχιστον για τις γυναίκες αυτό και για τα κοινωνικά οικονομικά εργασιακά θέματα όπως επίσης και για θέματα εκπροσώπησης. Ζητάω λοιπόν να επαγρυπνούν ε, τα ευρωπαϊκά όργανα, ιδιαίτερα προσεκτικό και με ιδιαίτερο θάρρος και δυναμικά να προχωρούν όπως ε, γίνεται και μέσω της πρωτοβουλίας αυτής. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες και εξουσίες. Θα πρέπει ιδιαίτερα να επιμείνουμε σε αυτό, για την εξουσία, ναι, είναι πολίτες ε, με τη λιγότερη δύναμη οι γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Χάρτα των Δικαιωμάτων, όπως επίσης και σε διάφορα ε, άλλα που έχουν θεσπιστεί. Θα πρέπει να υπάρξουν ακόμα περισσότερα μέτρα για ειδικά θετικά υπέρ των γυναικών για να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα. Ε, δεν μπορούμε να πούμε να τα παρνηθούμε αυτά. Η Ιταλία έχει μια χαμηλότερη ακόμα γυναική εκπροσώπηση. Και ορισμένες χώρες, στην περίπτωσή τους, που υιοθέτησαν ε, νόμους όπως η Γαλλία, το Βέλγιο θα μπορούσαν για μας να αποτελούν ένα φαρό, ένα σημείο αναφοράς για τη μάχη αυτή των γυναικών και θα πρέπει όλοι μας να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια, ακόμα περισσότερη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή και ως όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα οποία απευθύνω και τη σχετική πρόσκληση για να ανταποκριθούν. Ευχαριστώ. Grazie, ε, ε, ε, Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Μπέρα Μπεατρίτσε Λορεντσίνα από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα συνάδελφοι και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη δουλειά της, για τις προσπάθειές της και για μας και για την Ιταλία είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα ε, καθημερινά και να εμπιστοποιούμε τον κόσμο. Σήμερα μιλάμε για το μείζον θέμα. Την εκπροσώπηση των γυναικών και τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον αριθμό των γυναικών που εκλέγονται στα όργανα απόφασης και σε τοπικό επίπεδο, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό. Στην Ιταλία, το, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος σε ό,τι αφορά το, τη Βουλή, το Κοινοβούλιο, δηλαδή ε, με συγκεκριμένους ε, καταλόγους ε, βελτίωσε την εκπροσώπηση των γυναικών. Σήμερα όμως αντιμετωπίζουμε ένα, μια νέα πρόκληση τις ευρωπαϊκές εκλογές με ένα εκλογικό σύστημα αναλογικό, καθαρά αναλογικό. Σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να υλοποιήσουμε το στόχο της ίσης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών. Ε, μιλάω για την Ιταλία, αλλά φαντάζομαι ισχύει και για άλλε χώρε. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη η δουλειά που μπορεί να κάνει η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση ε, των πληθυσμών μα είναι πάρα πολύ σημαντική. Κάτι άλλο. Ε, μας ανησυχεί πάρα πολύ το θέμα, το... Μας απασχόληση. πάρα πολύ το θέμα της ε, γυναικής ε, απασχόλησης. Ε, υπάρχει οικονομική κρίση, προσπαθούμε να δουλέψουμε σε... να φτιάξουμε ένα χάρτη για την απασχολησιμότητα των γυναικών, για την ε, πρόσβαση των θέσεων εργασία, όλων των θέσεων εργασία ε, από τις γυναίκες. Φοβάμαι όμως ότι το τίμα θα είναι ψηλό από τους, ε, λόγω της κρίσης ε, που θα πληρώσουν οι νέοι και οι γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε για οικονομικά μέτρα κατά της κρίσης, προκειμένου να αποφύγουμε ε, να, μην, να χάνονται θέσεις απασχόλησης και κυρίως θέσεις απασχόλησης για τις γυναίκες. Κυρίως ε, θα ήθελα να τονίσω και ένα άλλο θέμα, ε, το θέμα τη βία κατά των γυναικών. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπρασπιστούμε τη γυναίκα από πολλέ απόψει. Και σε κοινωνικό και σε πολιτικό και σε πολιτιστικό, αλλά και σε ανθρώπινο. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο η εκπρόσωπο από την Κύπρο, Τη επιτροπή Ισότιμων Ευκαιριών, Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η κυρία Κουκουμά, Ε, από μέρου τη επιτροπή Ισότιμων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Κυπριακή Δημοκρατία, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση και την οργάνωση τη εκδήλωση αυτή. Η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων συνεχίζει να υφίσταται και εκτείνεται σε όλο το φάσμα της δημόσιας ζωής είτε αφορά την, στην εργασία, τις ευκαιρίες ανέλυξης και τη μισθοδοσία, είτε αφορά την πολιτική και τις ευκαιρίες συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στην περίπτωση της Κύπρου, ενώ πέραν του 51% των ψηφοφόρων στη χώρα είναι γυναίκες, το γυναικείο φύλλο εκπροσωπείται στη Βουλή με ποσοστό 8%, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο η Κύπρια γυναίκα είναι απούσα. Παρ' όλα αυτά, η εισαγωγή ποσοστώσεων ω έστω προσωρινό μέτρο εξάλληψη τη ανισότητα δεν μα βρίσκει σύμφωνου. Η συμμετοχή των γυναικών στι εκλογέ και στα σώματα λήψη αποφάσεων μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο εάν υιοθετηθούν μέτρα με ουσιαστικά και αηφόρα αποτελέσματα. Και εδώ είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει τέτοιε πολιτικέ που να στηρίζουν τη γυναίκα. Παραπέρα, η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια η εκλογή γυναικών στα διάφορα αξιώματα και σώματα λήψη αποφάσεων πρέπει να εντάσσεται μέσα στη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμιση τη συμμετοχή τη γυναίκα γενικά στην πολιτική ζωή και στην άνοδο τη πολιτικοποίηση στο γυναικών σε πλατιά βάση. Γιατί δεν υπάρχει αντρική και γυναικεία πολιτική. Γιατί γυναίκε πολιτικοί δεν έχουν προωθήσει πολιτικέ που να στηρίζουν πραγματικά τι γυναίκε και να εμπεδώνουν την ειρήνη. Και σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα με την ευκαιρία που όπως έχετε ανακοινώσει βρίσκεται εδώ η Τουρκάλα Υπουργό ε, για τα Δικαιώματα της Γυναίκας να την καλέσω να στηρίξει την κυβέρνηση, να, να, να ασκήσει πιέσεις έτσι που η κυβέρνηση της χώρας της να σταθεί θετικά και να στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται στην Κύπρο για διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Εδώ είναι η θέση της γυναίκας και εδώ είναι η ώρα για να αποδείξει αν πράγματι σαν γυναίκα έχει διαφορετική πολιτική. Ευχαριστώ. Ε, e, e, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Μάλτας, μέλος της Επιτροπής των Κοινωνικών Θεμάτων, κυρία Ζήστην Τερουάνο, παρακαλώ. Thank you, Madam Chairman. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε η εκπροσώπηση των γυναικών, ε, η ίση εκπροσώπηση των γυναικών αναγνωρίζεται από όλους. Αλλά συχνά τα προβλήματα παραμένουν ε, στις διάφορες κοινοβουλευτικές θητείες. Νομίζω ότι είναι και καινή ώρα να αρχίσουμε να συζητάμε για τις ποσοστώσεις, για να ε, καλυφθεί αυτό το έλλειμμα της γυναικείας εκπροσώπησης και στις Εθνικές Βουλές και στο, στην Ευρωβουλή. Όμως δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνο στη θετική διάκριση, γιατί μπορεί ναι, να, φτάσουμε τα νούμερα που θέλουμε, αλλά να έχουμε πρόβλημα με την ποιότητα. Νομίζω ότι οι γυναίκες θα πρέπει να αξιοποιηθούν όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο. Οι γυναίκες αποκλείται να ασχοληθούν και να διαφερθούν με την πολιτική, αν δεν ε, καλύψουμε και δεν ε, ανατρέψουμε όλες τις, ε, όλα τα προβλήματα που παραμένουν ε, εις βάρος των γυναικών σε όλους τους τομείς. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσα μισθοδοτικά δικαιώματα θα, για άνδρες και γυναίκες. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βία στο σπίτι, ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και, στην, τις ευκαιρίες, και ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Έχουμε κάνει πολλά υπέρ των γυναικών, αλλά υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά προβλήματα. Πολλές γυναίκες παλεύουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα λοιπόν πρέπει να τις υποστηρίζουμε ε, εναντίον όλων των μορφών ε, διάκριση Την ε, παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών κάθε γυναίκα στη περιμένει από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προστατεύσουν τα δικαιώματά της και τη ζωή της. Αν δεν υλοποιήσουμε αυτές τις προδοκίες, αποκλείεται οι γυναίκες να αισθανθούν εμπιστοσύνη για να ασχοληθούν ε, με την πολιτική σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο. Το να είναι κανείς πολιτικός χρειάζεται μεγάλη αντοχή, μεγάλη αποφασιστικότητα. Επομένως, ε, θα ήθελα να απευθύνω ένα κάλεσμα στις υποψήφιες ε, γυναίκες για τις ευρωεκλογές. Τους εύχομαι καλή επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και ελπίζω ότι περισσότερες γυναίκες θα επιλέξουν περισσότερες γυναίκες. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουλευτά. Και τώρα, με μεγάλη μου χαρά, μπορώ να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Σλοβακικής Βουλής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας απευθύνω μερικά λόγια εξ ονόματος της ε, Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών του, της ε, Βουλής της Σλοβακίας. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που δόθηκε με την ε, διάσκεψη αυτή να σας συναντήσουμε και να μιλήσουμε για τα θέματα των γυναικών στη Σλοβακία, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ε, για την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ανεξαρτήτως του πόσο αγωνιζόμαστε εμείς, τα αριθμητικά στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Και θέλουμε τελείως διαφορετική κατάσταση να εξασφαλίσουμε. τρεις γυναίκες θέλουμε να εκλέγονται, θέλουμε να στρατεύονται και να αγωνίζονται οι γυναίκες στον πολιτικό βίο, διότι δεν υπάρχουν όροι προϋποθέσεις ε, επαρκής που να επιτρέπουν στη γυναίκα στη Σλοβακία να συνδυάζει τον επαγγελματικό της ρόλο πολιτικό ενδεχομένως με τον οικογενειακό ρόλο της. Έχουμε ενώπιον μας ιστορική σημασία εκλογές, μια πολύ ισχυρή υποψήφιο στον, ε, για τη θέση της, ε, του, της Προέδρου στην Σλοβακική Δημοκρατία ε, μία θέση η οποία φαίνεται ότι ίσως να κερδιθεί από κάποια γυναίκα τελικά. Γιατί εάν ε, αποφασίσουν περισσότερες γυναίκες να προσφέρουν την ψήφο τους υποψήφιο γυναίκα, τότε ασφαλώς θα εκλεγεί γυναίκα. Η κυρία αυτή λοιπόν, ε, εάν εκλεγεί, ίσως μπορέσει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, να γυρίσει μια νέα σελίδα στην ε, ιστορία της γυναίκας στη Σλοβακία, το ρόλο της και την αποδοχή της από το δημόσιο βίο. Θα ήθελα να παρακαλέσω να ευχηθούμε όλοι από κοινού καλή επιτυχία στην κυρία αυτή, ώστε να έχουμε από τις 5 Απριλίου και μετά γυναίκα πρόεδρο της Σλοβακίας, η πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ας ακούσουμε την κυρία Βιπιάννα Βιτσοβάσκοβα, η οποία είναι η εκπρόσωπος της πρώην Δημοκρατία Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, λέγομαι Βουπόφσκα από την ΦΥΡΟΜ. Ε, εκπροσωπώ την, εκπροσωπή, την Επιτροπή Ίσης Εκπροσώπησης Ανδρών και Γυναικών. Ε, ανήκω στο Πράσινο Κόμμα. Ε, συγχαρητήρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή τη διάσκεψη. Στην Μακεδονία, συγγνώμη, όχι στη ΦΥΡΟΜ. Ε, έχουμε αυξήσει πέντε φορές τα τελευταία έξι χρόνια την ποσότητα των γυναικών το ποσοστό γυναικών, από το 6% στο 31%. Έχουμε φτάσει περίπου στα ποσοστά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαστε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο ίσοι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο που προασπίζει τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μου δεν ε, σταματάμε μπροστά σε κανένα σύνορο, πολιτικό, θρησκευτικό, φιλετικό. Ε, και με αυτόν τον τρόπο ε, συμμετέχουμε στην αύξηση της συνοχής της χώρας μας. προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερα νούμερα γυναικών στην πολιτική, αλλά όχι μόνο αυτό. είμαστε και υπάρχει της ποιότητας για να προσπιζόμαστε τα δικαιώματα των γυναικών στην κοινωνία γενικά. Ε, Μακεδόνισες γυναίκες ε, συμμετέχουν σε αυτή την εκστρατεία ε, γυναίκες στην πολιτική 50-50. Και έχουμε ε, συγκεντρώσει μέχρι στιγμής χίλιες υπογραφές. Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Υψίστας Ευκαιρίας ανακοινώθηκε αυτή η εκστρατεία. Πρέπει να πω όμω ότι μόνο μαζί με τους άντρες, άντρες και γυναίκες μαζί, θα δημιουργήσουμε μια διαφορετική πραγματικότητα, ε, μια πραγματικότητα με ισοτιμία για του άντρε και τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Κυρία εκπρόσωπο της Μακεδονίας και τώρα στο τέλος της συζήτησης μπορούμε να ακούσουμε την εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ ξεκινώντας για την οργάνωση αυτής της συνάντησης ε, και μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, το οποίο εγώ εκπροσωπώ σήμερα ειδικότερα για την Επιτροπή για την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Θα ήθελα να εκφράσω μια άποψη προς την κατεύθυνση τώρα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητώμε για τις γυναίκες και για το επίδο εκπροσώπησης των, ε, στην λήψη αποφάσεων. Σημαντικό είναι γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού και των κρατών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης και η συμμετοχή των γυναικών στα όργανα που λαμβάνονται αποφάσεις δεν είναι η πραγματικ... ο αριθμός τους με τον πραγματικό αριθμό Τα 27 από τα κράτη ασχολούν, απασχολούν περισσότερο, λιγότερες από 40 40% των θέσεων που είναι ο ελάχιστο, το ελάχιστο ποσοστό που υποδεικνύει το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν αρκετή εκπροσώπηση γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων και εδώ στο ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης εκφράζεται το 78% από συμμετέχουν από εθνικά κοινοβούλια, αριστερών ε, από εθνικούς οργανισμούς, είναι γυναίκες μόνο το 22% είναι γυναίκες. Ε, όταν λέμε ότι θέλουμε ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει αυτή την ισότητα για από τη στιγμή που δεν είναι το ποστό γυναικών σύμφωνα με το ποσοστό στο αριθμητικό. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και για κοινωνική δικαιοσύνη, για παρόμοιους λόγους. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε ενέργειες που να διευκολύνουν τις γυναίκες να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Και μετά πως έχουν γίνει το 1995 μέσω της πλατφόρμας της τέταρτης παγκόσμιας συνδιάσκεψης γυναικών στο Πεκίνο που αναφέρθηκε και όσο ποτέ η ανάγκη συμμετοχής των γυναικών είναι από εκείνα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα επειδή δεν έχουν επιτευχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως τώρα τελευταία αναγνωρίστηκε και από την Γενοφική ε, συνέλευση τα κόμματα τα πολιτικά έχουν ιδιαίτερα ευθύνη τώρα που θα πρέπει να προωθήσουν τις γυναίκες ε, σε αυτές τις υψηλές πολιτικές θέσεις ε, και στα πολιτικά κόμματα στις θέσεις λήψης αποφάσεων. Κυρίες και κύριοι, για αυτό το λόγο η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, θέλησε να συγχαρεί τα όσα έχουν γίνει από τα πολιτικά κόμματα και έχουν επιτρέψει τη βελτίωση την ιδιαίτερη της συμμετοχής των γυναικών σε αυτές τις συνελεύσεις, στα πολιτικά κόμματα και στα εκτελεστικά όργανα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, λοιπόν, ε, μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που γίνονται παρόμοιες ενέργειες σε αυτά τα πολιτικά κόμματα, θα ήθελα από τη στιγμή που έχουν σημειωθεί παρόμοια βήματα να μας τα ανακοινώνετε και ακριβώς για να μπορέσουν να επιβραβευθούν από το βραβείο περισσότητος που έχουμε θεσπίσει στη συνέλευσή μας και μέχρι τις 1η Ιουνίου του 2009 υπάρχει προθεσμία για την υποβολή υποψηφιών υποψηφιότητων για το βραβείο αυτό είναι ένα έργο όλων μας και στα πολιτικά μας κόμματα στα οποία ανήκουμε, τα οποία εκπροσωπούμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε ώστε οι γυναίκες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης, τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες σε όλες τις θέσεις και εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις. Να υποστηρίξω χωρίς καμία επιφύλαξη την Επιτροπή των Ευκαιριών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Και σίγουρα εμπιστεύομαι την στενή αυτή συνεργασία γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από κοινού για να πετύχουμε το στόχο μας που ο στόχος μας είναι η βελτίωση της συμμετοχή γυναικών στις εκλεγμένες αυτές συνελεύσεις. Όσο ποτέ σήμερα θα πρέπει να ακουστεί η φωνή των γυναικών και στα όργανα λήψεων αποφάσεων. Έτσι θα έχουμε ένα δικαιότερο κόσμο με ίσες ευκαιρίες και να μην είναι κάτι το τοπικό να αποτελέσει πραγματικότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Ευχαριστώ θερμά την εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης και τώρα παρακαλώ να προχωρήσουμε με τη συζήτησή μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την διοργανική συνεργασία με τις συναδέλφους βουλευτές για να ακούσουμε πρώτη την κυρία Αστρίτ Λούλινγκ, βουλευτή από το Λουξεμβούργο, ευρωβουλευτή από το Λουξεμβούργο, η οποία είναι παρούσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 30, αν το πιστεύετε, συναπτά έτη. Η κυρία Λούλινγκ είναι κοσμήτωρα, έχει πολλές ευθύνες ε, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως μπορεί να μας εξηγήσει πώς μπορεί κανείς και βέβαια να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και πώς μπορεί να μείνει τόσο πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Λούλινγκ, έχετε το λόγο. Ε, euh, Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα διαπιστώσατε ίσως στην παρουσίαση της κυρίας Πρόεδρου ότι η ηλικία μου είναι αυτή που μου εξασφαλίζει το προνόμιο να σας ομιλώ σήμερα εδώ ως πρεσβυτέρα. Επισημαίνω πάντως ότι δεν είμαι η πιο ηλικιωμένη του Κοινοβουλίου. Άντρας έχει την τιμή αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε ακόμη έναν-δύο κυρίους πιο ε, ηλικιωμένους από μένα. Γυναίκα όμως η πιο ηλικιωμένη είμαι εγώ. Ή, αν το θέλετε να το πω διαφορετικά, το παλαιότερο μέλος, ο παλαιότερος βουλευτής. Από τους 785 όμως είμαι η μόνη η οποία ήταν μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης πριν από τις άμεσες καθολικές εκλογές του 1979 γιατί το 65 ήδη ήμουνα τότε το νεότερο μέλος και μακράν νεότερο και ίσως από, τους, από τις λίγες γυναίκες ήταν πολλοί οι άντρες και πιο ηλικιωμένοι από μένα 10, 20, 30 χρόνια περισσότερο από μένα είχε ο καθένας τους και μάλιστα ε, χάθηκαν με τον ένα τον άλλο τρόπο από το προσκήνιο. Εν πάση περιπτώσει όμως αφού ξεκίνησα εγώ τότε η νεότερη στην ε, συνέλευση εκείνη, α είμαι μια φορά και η πιο ηλικιωμένη. Να δούμε τώρα τον επόμενο Ιούνιο, εάν θα μείνω για να διεκδικήσω και την ηλικία. Η Αν Μαρή Ρέγκερ, Γερμανίδα, βουλευτής που τη γνώριζα από την εποχή της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όταν ήμουνα κοπέλα, άλλαξε βέβαια πολλά πράγματα από τότε, μου είχε πει μια μέρα, Άστρετ, ξέρεις, εμείς εδώ οι γυναίκες, Μόνο πατώντας πάνω σε πτώματα ανδρών μπορούμε να έρθουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Αστεϊσμός φυσικά, αλλά ταυτόχρονα και μία σκέψη η οποία από την πρώτη εκείνη στη συνέχεια πρόεδρο του γερμανικού Bundestag και μορφή μεγάλη της γερμανικής ε, πολιτικής μπορεί βέβαια να μας ε, κάνει να, χαμογελάμε πλην όμως είναι και πολύ αποκαλυπτική ως παρατήρηση. Πολλές είμαστε αυτές που είδαμε αυτό ακριβώς τον όρο να υλοποιείται. Η Άρμαντε Διρέγκερ δεν θα μπορούσε στη δική μου συγκεκριμένα περίπτωση να είχε προβλέψει πιο εύστοχα όταν στις, στις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές του 1964 ήμουν η μόνη γυναίκα υποψήφιος του κόμματός μου για ολόκληρη τη χώρα του Λουξεμβούργου. Κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσα τη γυναίκα άλοθη των εκλογών εκείνων. Κακό δεν ήταν φυσικά, γιατί τελικά εξελέγει τρίτη, μάλλον ορίστηκα τρίτη αναπληρωματική στον κατάλογό μου, στην εκλογική μου περιφέρεια και επισημαίνω ότι στο Λουξεμβούργο δεν προσδιορίζει το κόμμα την τάξη της εγγραφής στον στην εκλογική λίστα, αλλά οι ψηφοφόροι, τα μέλη καλύτερα του κόμματος, με την ψήφο τους. Φυσικά, το εάν θα συμπεριληφθεί κάποιος στον κατάλογο, το ορίζει το κόμμα, αλλά ο ψηφοφόρος, η βάση, είναι εκείνη η οποία ορίζει το, τη σειρά την εκλόγιμη και βέβαια πρέπει να σημειώσω ότι εγώ πάντοτε καλύτερα τα πήγαινα με το λαό παρά με τα κόμματα. Τα κόμματα στα οποία ε, ήμουν μέχρι τώρα σε αυτή τη βάση μπόρεσα να τα χειριστώ και να έχω σχέση μαζί τους. Σε βάση περιπτώσει όμως χάρη και στον θάνατο κάποιων ε, ε, ανδρών συναδέλφων μπόρεσα να βρεθώ το 1965 σε υψηλότερη θέση ε, το 1965 και να βρεθώ σε εκλόγιμη θέση, δεύτερη θέση συγκεκριμένα το 1965, μόνη γυναίκα στο Λουξεμβούργο, στο Κοινοβούλιο του Κοινοβουλίου. Για χρόνια δεν υπήρχε γυναίκα στο Κοινοβούλιο, ούτε μια γυναίκα στους, γενικά στη δημόσια διοίκηση δεν υπήρχε, για να σας εξηγήσω, ούτε τουαλέτες γυναικείες δεν υπήρχαν στα κτίρια του Κοινοβουλίου μας τότε. Έτσι λοιπόν ο κόσμος της πολιτικής ήταν τελείως αρενοπός το 65 εκείνο όπου γίνομαι ταυτόχρονα εθνική βουλευτής και μέλος της συνέλευσης του, που έγινε μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γυναίκες λοιπόν και οι άντρες είχαν κάτι μεγάλα πουρα που κάπνιζαν στη συνεδριάση των επιτροπών. Μάλιστα πουρα που τους τα προσέφερε δωρεάν ε, το κοινοβούλιο. Περνούσαν οι κλητήρες του κοινοβουλίου με τα κουτιά και τους σερβίραν πουρα στη διάρκεια των συνεδριάσεων. Ομολογώ πάντως ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ ε, άβολα που θα ήμουν ε, μόνη γυναίκα μεταξύ ανδρών, γιατί είχα την τύχη στην οικογένειά μου να είμαι το μόνο κορίτσι με τρία μεγάλα γόρια. Και όπως καταλαβαίνετε στις κλωτσοπατινάδες θα πήγαινα πολύ καλά μαζί τους. Έτσι ήμουν έτοιμη και για την αντιπαράθεση στο λουξεμβουργιανό κοινοβούλιο όταν βρέθηκα μόνη μου και ο πρόεδρος τότε του κοινοβουλίου, μεγάλος πολιτικός του Λουξεμβούργου, ο κύριος Βέρνερ, μου είπε «Μα Άστριτ, μόνη σου με τόσους άντρες δεν φοβάσαι». Η απάντησή μου ήταν «Ναι, «Πρόεδρε, εγώ είχα τρεις αδελφούς μεγαλύτερους, δεν φοβάμαι τίποτα». Όντως λοιπόν ο αγώνας των γυναικών μέσα στην πολιτική είναι μακρύς και σκληρός τίποτε να μας προσφέρετε δωρεάν και γι' αυτό οφείλουμε πιστεύω πολύ μεγάλο φόρο τιμής σε όλες εκείνες και εκείνους βέβαια που μας στηρίζουν στον αγώνα αυτών Ταυτόχρονα στην πορεία αυτήν που άλλωστε δεν έχει ακόμα καταλήξει, δεν έχει φτάσει σε δικαίωση, θα πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα έναν αγώνα κατά των αδικιών. Κυρίε και κύριοι, σε αυτά που κάνουμε δεν είμαι διατεθειμένη να δώσω χαρακτηρισμό μανιχαϊστικό το, κακό αγωνίστε, το καλό αγωνίστε κατά του καλού. το καλό κατά του κακού. Γιατί ευθύνη έχει και η γυναίκα να αναλαμβάνει τις καλές, τις σωστές επιλογές για να προαγάγει την ισότητα. Αντί λοιπόν για να διαμαρτυρόμαστε και να παραπονιόμαστε, ας γυρίσουμε το βλέμμα πριν πίσω και ας προσμετρήσουμε το δρόμο που έχουμε διανύσει όλο αυτό το διάστημα με το 30% τώρα των γυναικών ευρωβουλε... των ευρωβουλευτών που είναι γυναίκες αυτή τη στιγμή για μας το Λουξεμβούργο, χώρα κατ' μικρότερη από τη Μάλτα, το ποσοστό συμμετοχής ανδρών και γυναικών βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απόλυτα ισορροπημένο. Τρει άνδρες, τρει γυναίκε. Είμαστε έξι συνολικά. Μάλιστα στο Λουξεμβούργο είχε εκφραστεί ο φόβο ότι θα ήταν περισσότερε οι γυναίκε από ότι οι άντρε ε, που θα προέκυπταν ε, ω ευρωβουλευτέ στι τελευταίε εκλογέ. Πριν από λίγο ο πρόεδρο Πέτερινγκ σα είπε Πόσε είναι οι γυναίκε οι οποίες έχουν ε, θέσει ευθύνη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ μπορώ να σα εξηγήσω ότι μπορεί να μην είμαστε παρά το 1 τρίτο οι γυναίκε ευρωβουλευτές μεταξύ των 785, πλην όμως πολλέ είμαστε εκείνες οι οποίες με τη δουλειά μας, με την επιμονή μας, με την ε, επιμέλειά μας και τις ικανότητές μας μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χάσμα. Και από την άλλη δεν είναι και λίγοι οι άντρες οι οποίοι έχουν ε, πολύ ε, χαλαρή θα έλεγα παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μάλιστα και δημοσία στις εφημερίδες ακόμη δηλώνουν ότι δεν ασχολούνται με την κοινοβουλευτική εργασία και δεν μπαίνουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές κτλ. που όμως για άλλους λόγους έχουν πολύ μεγάλη προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί είναι κυρίες και κύριοι οι άντρες οι οποίοι κάνουν κακό στη δουλειά μας και που κάνουν κακό στα δικαιώματα των γυναικών ή εκείνοι οι οποίοι έστω και με καλές προθέσεις δεν ε, σταματούν να μας δημιουργούν προβλήματα και να μας οδηγούν σε αντιπαραθέσεις και κυρίως μέσα στην Επιτροπή των Γυναικών με των δικαιωμάτων των γυναικών με ακραίες ακόμη διεκδικήσεις μερικές φορές προσπαθώντας τις γυναίκες να τις θέσουν σε καθεστώς επιτροπίας να τις προστατεύουν πάση θυσία οι πάντες αντί να τις αφήνουν να αναπτύξουν τις δυνατότητες του ελεύθερου προσπαθούν να του να τους επιβάλλουν μόνο και μόνο για λόγους κάποιες προβολής αρμοδιότητες και ευθύνες σε διάφορους τομείς. Έτσι λοιπόν και για να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο θα πρέπει να, κάνουν, να γίνουν οι σωστές επιλογές, οι, σωστές, ε, οι σωστοί προσανατολισμοί. Και αυτό πρέπει να το κάνουν οι γυναίκες πάνω απ' όλα. Στις ποσοστώσεις πίνε. Εγώ πιστεύω ότι η υποχρεωτική ποσόστοση, που άλλωστε έχει και το δικό μου το κόμμα τώρα, η ποσόστοση είναι το πω διαφορετικά υποχρεωτική ή μη, έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ενισχύσει την ε, εκπροσώπηση των γυναικών σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Πλην όμως εγώ δεν είμαι δογματική, δεν διεκδικώ μια μαξιμαλιστική πολιτική στην υπόθεση αυτή. Και όταν βλέπω πόσες ζημιές μπορεί να, έχει προκαλέσει η υποχρεωτική εναλλαγή ανδρών και γυναικών στον κατάλογο των των υποψηφίων ε, για τις ευρωεκλογές, κυρίως σε ορισμένα κόμματα, θα έλεγα ότι μερικοί το τραβάνε υπερβολικά το σκηνή. Και ερωτώ, γιατί να μην έχουμε έναν καλό υποψήφιο, γιατί δηλαδή να στερηθούμε ένα καλό υποψήφιο και το κριτήριό μας είναι μόνο σε ποιο φίλο ανήκει κανείς, αν είναι το καλό ή το κακό φίλο. Αυτό. Δεύτερον, στις γυναίκες οι οποίες θέλουν να αναλάβουν δραστηριότητα στην πολιτική, συνιστώ πάντοτε τις αποφάσεις να τις παίρνουν με σοφροσύνη. Κυρίε και κύριοι, μην επιμένετε πάντοτε να ε, προσανατολίζεστε προ ε, τι υπηρεσίε τη κοινωνική ιατροφαρμακευτική. Περάστε και στου άλλου τομεί, αυτού που θεωρούνται ότι είναι τα φρούρια των ανδρών, οικονομία, ε, πολιτική, χρηματοπιστωτικά κτλ. Κάποιο μου λέει ότι πρέπει να τελειώνω, δεν ξέρω γιατί. Πώ είναι δυνατόν να σταματήσω να μιλάω. Αν δεν σα πω ότι Για να καταλήξω ότι το να βρισκόμαστε, το να ζούμε σε έναν κόσμο ανδρών, το να ζω εγώ σε έναν κόσμο ανδρών, εμένα δεν μου δημιούργησε πρόβλημα, δεν με έφερε ποτέ σε μηχανία. Του αντίον μάλλον. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψω κιόλας να πω ότι στη μακρά μου πολιτική σταδιοδρομία διανύω τώρα τη 16η μου προεκλογική περίοδο μαζί με εθνικές βέβαια και κοινοβουλευτικές ε, εκλογές, ευρωεκλογές υπολογίζοντας εγώ λοιπόν σε όλη μου αυτή την ε, σταδιοδρομία προβλήματα δεν είχα ποτέ με τους ευφυείς άνδρες συναδέλφους πολιτικούς. Μόνο με κάτι... Ε, με κάτι φαλοκράτες ανόητους είχα αντιπαραθέσεις και προκλήσεις ε, και προβλήματα και πάνω απ' όλα με ορισμένες γυναίκες πολύ πιο ανόητες, διότι δυστυχώς η χειρότερο, ο χειρότερος εχθρός της γυναίκας, από ό,τι διαπιστώνω, είναι η ίδια η γυναίκα σε ορισμένες περιπτώσεις. Με εξαιρέσεις βέβαια. Αλλά έχω πολλές εμπειρίες που θα μπορούσα να σας περιγράψω, αν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και ίσω πολιτικά να μην θεωρείτε κομψό. Αλλά πάντω ήθελα να σα εκφράσω τι εμπειρίε μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Λούλιν. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε και για τις επόμενες βέβαια ευρωεκλογέ. Και τώρα, ας λάβει παρακαλώ το λόγο η κυρία Ζήτα Κουρμάη, ευρωβουλευτής από την Ουγγαρία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της ε, ισότητας των ευκαιριών. Σήμερα η κυρία Κουρμάη θα μας ε, μιλήσει και για τις άτυπες σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το διοργανικό δίκτυο που έχει, του οποίου ηγείται. Κυρία Κουρμά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, συμπατριώτες και συμπατριώτησές μου από την Ουγγαρία και από την ε, Ουγγρική Βουλή. Έχουμε έναν άντρα και μία γυναίκα που εκπροσωπεί εδώ την Ουγγαρία. Θα ήθελα παρόλα αυτά να καλωσορίσω εξίσου θερμά και όλους τους υπόλοιπους ανεξάρτητος φίλου. Φυσικά θα συνεχίσω στα αγγλικά. Γιατί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μήνυμα περνάει μόνο αν μιλάει κανείς αγγλικά. Με μεγάλη τιμή είμαι εδώ μπροστά σας, σε αυτή την εκδήλωση της Επιτροπής Γυναικών. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτή την ε, θαυμάσια εκστρατεία για την ε, ίση εκπροσώπηση 50-50 άνδρες και γυναίκες. Ε, οι περισσότεροι επίτροποι υπέγραψαν, ο κ. Μπαρόσο υπέγραψε, αλλά ο κ. Πέτερν δεν έχει υπογράψει. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Αν είναι μια βασική αρχή ισότητα ανδρών και γυναικών, ε, στις, είναι πολύ σημαντική επίσης για μια δημοκρατία και ίση συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, στην κοινωνία κτλ. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος πρέπει να υπογράψει αυτή την ε, προσπάθεια. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν συμφωνεί ο πρόεδρος του ε, Κοινοβουλίου ότι χρειαζόμαστε 50% άνδρες και 50% γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχει ένα πράγμα με το οποίο Δυστυχώ, δεν θα συμφωνήσω με την προηγούμενη ομιλήτρια. Φυσικά θέλω οι καλύτεροι να προχωρούν. Αλλά γιατί ζητάμε πάντα τι γυναίκε να είναι καλύτερε και δεν ζητάμε το ίδιο και για του άντρε. Εγώ θέλω λοιπόν να υπάρχει διπλή ποσότητα και για άντρε και γυναίκε. Γιατί α τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Κοιτάξτε αυτά που είπε η συνάδελφο από την Μακεδονία. Η Task Force για, το, για τα δύο φύλλα έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Πραγματικά, ε, συγχαρητήρια, θέλουμε να σας βοηθήσουμε στην περιοχή σας για να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Αυτό το δίκτυο γυναικών είναι πάρα πολύ ισχυρό και βοηθάει την όλη προσπάθεια. Οι ποσοστώσεις ξέρω ότι είναι ένα μόνο εργαλείο, αλλά βοηθάει σίγουρα την εκπροσώπηση των γυναικών και εφόσον τη βοηθάει, το θέλω αυτό το εργαλείο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε 30% γυναίκες. Οι περισσότερες είναι πράσινες. 47% από το 30% είναι γυναίκες. Εν συνεχεία, φιλελεύθεροι. Φυσικά, μόνο 11% έχει το ΟΕΝ. Ε, και το ΕΛΚ 23% γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν προωθούμε τις πολιτικές ε, και στις ευρωπαϊκές εκλογές να αποδεικνύουμε ότι κάνουμε κάτι για το 52% του παγκόσμιου πληθυσμού. Υπάρχει μάλιστα και ένα κόμμα το οποίο τι πρέπει να κάνουμε για την ισότητα άνδρων και γυναικών. Ετοιμάσαμε αυτό το μανιφέστο, το οποίο συζητήσαμε επί ένα χρόνο, ε, με τους απλούς πολίτες. Ακούστε τι είπε η κυρία Βάλστρομ. Θα πρέπει να μιλήσουμε στον απλό άνθρωπο, στον δρόμο. Θα πρέπει να κατεβούμε στον δρόμο, στις πλατείες. Ε, Υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ε, γυναικών πιστεύουν ότι η πολιτική, και οι άντρες το πιστεύουν βέβαια, ότι η πολιτική κυριαρχείται από τους άντρες. Μόνο αν ένα κόμμα έχει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για την ισότητα ανδρών των γυναικών, μόνο τότε μπορεί να πείσει ότι προωθεί τα ε, δικαιώματα των γυναικών. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, πολύ περήφανη ε, από τη δουλειά που κάναμε και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρω ότι δεν με αγαπούν οι μεταφραστές και οι διερμηνείς γιατί μιλάω πολύ γρήγορα, αλλά τέλος πάντων. Είδατε τι έγινε στις εκλογές ε, και στα δημοψηφίσματα στην ε, Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιρλανδία. Οι γυναίκες ε, θέλησαν να πούν όχι στην Ευρώπη. Γι' αυτό αυτό το φυλάδιο. Η Ευρώπη μέσα από τα μάτια των γυναικών. Τώρα σήμερα βλέπουμε τι γίνεται, που έχουμε την κρίση. Ποιος προκάλεσε την κρίση. Ε, την προκάλεσαν εταιρείε τις οποίες τις διαχειρίζονται ποιος, οι άντρες ή οι γυναίκες, οι άντρες βέβαια. Επίσης κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, τι πιστεύουν ε, οι απλοί άνθρωποι για μας, τις γυναίκες. Οι γυναίκες στην πολιτική μπορεί να βοηθήσουν ε, να δώσουν μια προστιθέμενη αξία ε, στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Αυτό το πιστεύει μεγάλη ε, πλειοψηφία, παρά οι περισσότεροι που το πιστεύουν είναι γυναίκες παρά άντρες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τον κόσμο. Ε, χαίρομαι που η Τσέχα Υπουργό είναι εδώ μαζί μας. Συγγνώμη, ο Τσέχος υπουργό. Ε, θα ήθελα να μας πούνε όμως στην Τσεχία τι κάνανε για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εμείς ε, έχουμε βάλει σε εκλόκιμη θέση στον κατάλογο τρεις γυναίκες. Θα ήθελα ε, να γίνει έτσι ένας ανταγωνισμός μεταξύ μας, ένας αγώνας για το ποιος θα κάνει περισσότερα, ούτως ώστε να πετύχουμε την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά, πρέπει να μιλάμε για τις γυναίκες, πρέπει να μιλάμε για τις διακρίσεις που υφίστανται. Πολλές γυναίκες λένε ότι δεν αισθάνθηκαν ότι υφίστανται διακρίσεις λόγω του φίλου τους. Ε, καλό αυτό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι άντρες και γυναίκες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Δεν υπάρχει ίσω μισθό ανδρών και γυναικών για την ίδια δουλειά, όπω είπε και ο Πίτροπο Σπίτλερ. Γι' αυτό χαίρομαι αυτή την εκστρατεία που ξεκίνησε υπέρ τη ισοτιμία. Νομίζω ότι επειδή χρειαζόμαστε πολλά χρόνια για να κλείσουμε αυτό το χάσμα τη ψαλίδα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα, θα πρέπει να σκουμποθούμε τώρα. Επίση, κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον. Οι γυναίκε ενδιαφέρονται πιο πολύ για τα ευρωπαϊκά θέματα από του άντρε. Ενδιαφέρονται για αυτά που κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 39% των ε, γυναικών ευρωβουλευτών εκπονούν περισσότερες εκθέσεις από τους άρενες συναδέλφους τους. Μερικές φορές λοιπόν ε, είμαστε πράγματι καλύτερες από τους άντρες. Αυτά και δεν θέλω να μακρηγορήσω και θέλω να δώσω και λίγο χρόνο στην επόμενη ομιλήτρια. Αλλά τι θέλω να σας πω, ότι στην Ισπανία α πούμε, ο Σαπατέρο κάνει μια θαυμάσια δουλειά. Προώθησε γυναίκα υπουργό κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνης τη. Η Υπουργό Αμήνη ήταν έγκυο όταν με το πόστο τη. Μπράβο. Επίσης, ε, προσπαθούμε και εμείς ε, στην Ουγγαρία Πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες να, και να τις βοηθήσουμε κυρίως να συμφιλιώσουν εργασία και οικογενειακή ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Στακουρμάη για την παρέμβασή σας. Ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα πιο ουσιαστικό τμήμα της ορεινή μα συζήτηση που είχα άλλωστε προεξαγγείλει, είπα ότι είχαμε μία μελέτη αναθέσει για το σύστημα των ποσοστώσεων όπως εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Την, την έκθεση αυτή τη μελέτη την ανέλαβε και την εκπώνησε το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Γι' αυτό θα παρακαλέσω την καθηγήτρια κυρία Ντάλερουπ να μας κάνει πολύ σύντομα τα αποτελέσματα της ε, μελέτης αυτής. Παρακαλώ κυρία καθηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας, την Πρόεδρο, για την ε, πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω ενώπιον της σημαντικής αυτής διάσκεψης. Όπως υπόθηκε, αναλάβαμε τη διεξαγωγή μιας μελέτης για τα συστήματα των ποσοστών σε εκλογές στα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πρωτοκαθεδρία στην ισότητα και τις ποσοστώσεις. Πλην όμω ε, και από τα όσα άκουσα και εδώ, διαπιστώνουμε ότι πολλά γίνονται και πολλέ πρόοδοι σημειώνονται σιγά σιγά. Από τη μελέτη μα και εμεί διαπιστώνουμε ότι κάποιε χώρε έχουν ήδη κάποιο σύστημα ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσει νομίζω ότι έχουν ρόλο καταλητικό για την αλλαγή. Μπορεί κανεί να στάσετε κατά των ποσοστώσεων ή υπέρ αυτών. Αλλά πάντω διαπιστώνουμε ότι έχουν καταλητικό ρόλο στην εκπροσώπηση περισσότερων γυναικών. Και ερωτώ, και ίσως αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει ως ερωτηματικό. Ας προχωρήσουμε λοιπόν ιστορικά πίσω, το 40-50, στην πολιτική επικρατούσαν οι άντρες, οποιαδήποτε πολιτικό θεσμό εμφανίζονταν γυναίκες, ήταν μια πολύ σπάνια εξαίρεση. Και θα ακούσατε ίσως και ότι και στη δεκαετία του 60, όπως μας πει η κυρία Λούλη, το φαινόμενο ήταν λίγο πολύ ε, το ίδιο. Μπορεί να είχαν οι γυναίκες το δικαίωμα του εκλέγην ε, σε ορισμένες χώρες γύρω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήδη ε, κερδίσει, πλην όμως ήταν λίγες οι εκλεγόμενες πολιτικοί γυναίκες. Ήταν πολύ περιορισμένη λοιπόν η εκπροσώπησή τους. Πάντως, πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι πριν από 50 χρόνια δεν θεωρούνταν μη δημοκρατική μία ε, συνέλευση κοινοβουλευτική στην οποία απο, η οποία παρτίζονταν αποκλειστικά από άντρε. θεωρώ τον αυτονόητο ή φυσιολογικό το να είναι μόνο άντρε βουλευτέ σε ένα κοινοβούλιο, το να μην υπάρχει ούτε μια γυναίκα. Αντίστροφα, το δικαίωμα του εκλέγην ε, στην ε, Ελβετία δεν αναγνωρίστηκε μέχρι το 1971. Είδαμε εκεί πέρα να γίνονται τίποτε διαδηλώσει ή και έξω από την Ελβετία εναντίον αυτού του συστήματο. Όχι. Ήταν αυτονόητο δηλαδή ότι η γυναίκα θα βρίσκεται στο παρασκήνιο. Ε, ταυτόχρονα βλέπουμε όμως ότι δεν είναι δημοκρατικό ή δεν θεωρείται ως δημοκρατικό από ορισμένε γυναίκες ή άντρες το να μην υπάρχει εκπροσώπηση τουλάχιστον κατά 30% στη σήμερον εποχή των γυναικών. Τουλάχιστον κατά 30% ή και 40%. Ο στόχος λοιπόν που ε, ορίζεται τώρα, ενώ παλαιότερα ζητούσαμε να υπάρχουν περισσότερε γυναίκε στις εκλογές, στις ε, πολιτικές αναμετρήσεις, στην πολιτική ζωή, τώρα έχει μετατραπεί ο στόχος σε ισότιμη συμμετοχή. Ισορροπία 50% ο ένας 50% άλλος, ένα προς ένα σε ορισμένε περιπτώσει όπω το λόμπι των γυναικών κτλ. ή όπω η Επιτροπή του Αφρικανικού Κοινοβουλίου ε, που λέει τουλάχιστον 5%. Και να σα πω ότι πρόκειται για μια από τι πιο προοδευτικέ ε, και πιο, πιο αγωνιστικέ ε, οργανώσει και ενώσει που έχω συναντήσει. Άρα πλέον ο κανόνα είναι ότι η δημοκρατία χωρί ισότιμη συμμετοχή των φίλων δεν υπάρχει. Και ε, σημειώνω για να μην παρεξηγηθώ ότι η παρουσία των γυναικών δεν αποτελεί τη μόνη πηγή νομιμοποίηση φυσικά, ούτε ε, λύνει όλα τα προβλήματα η παρουσία των γυναικών σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Η υποεκπροσώπωση των γυναικών είναι όμω ένα από τα πολλά δημοκρατικά ελλείμματα που σημειώνονται και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η συμμετοχή των γυναικών δεν μπορεί να επιλύσει φυσικά όλα τα προβλήματα. Όμω αναπτύσσεται ένας νέος δημόσιος διάλογος. Αλλάζουμε ορολογία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μετακινούμαστε πιστεύω από την ιδέα ότι η ισότητα θα έρθει εξ ουρανού ή από μόνη τη, συν το χρόνο και νομίζω αυτό ήταν ίσως η, η ευρωπαϊκή νοοτροπία η οποία ε, για μένα θα μπορούσε να περιγραφεί ως ε, ε, σορευτική χρονοθυρίδα, δηλαδή ότι σιγά σιγά μπορούμε να περιμένουμε όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στο δημόσιο βίο και αυτή πια έχει εγκαταληφθεί ως νοοτροπία βλέπω σιγά σιγά αντιθέτω να υπάρχει ανησυχία, αμηχανία, ενόχληση ακόμη των, γυναικών, των γυναικών γιατί δεν εκπροσωπούνται επαρκώ. Και υπάρχει σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά η τάση να ανατραπεί αυτή η επικυριαρχία, η μονοκαθεδρία των ανδρών στον πολιτικό βιοστήριο. Τελευταίε δεκαετίε δεν πρέπει να σα πω ότι ε, εισάχθηκε, εισήχθη το σύστημα των ποσοστώσεων σε 50 χώρε στον κόσμο, μέσα στα συνταγματικά του κείμενα ακόμη, σύστημα ποσοστώσεων για τι εκλογέ. συγκεκριμένα 47 είναι οι χώρες ανά τον κόσμο που γνωρίζουν αυτή τη στιγμή συνταγματική ή νομοθετική διάταξη για τις εκλογές τους, για τα εκλογικά του συστήματα και άλλες 50 αυτές τις οποίες τα κόμματα έχουν εισαγάγει σύστημα ποσοστώσεων για την συμμετοχή στις λίστες των γυναικών. Αυτό δείχνει μια τεράστια αλλαγή φυσικά. Επίση, η, άλλη, η άλλη αλλαγή που σημειώνεται είναι ότι αντί να κατηγορούνται οι γυναίκε πλέον για τα δεινά αυτά, κατηγορούνται οι θεσμοί, τα όργανα. Και πρέπει να κοιτάξουμε φυσικά και πώ λειτουργεί ένα σύστημα. Εγώ είμαι Σκανδιναβή, ζω στη Σουηδία. Η Καταγωγή μου είναι δανική, από τη Δανία. Αυτό που κάναμε λοιπόν εμεί εκεί, οι γυναίκε, αυτό που έκαναν οι γυναίκε και πριν από μένα, ήταν ότι κάθισαν να δούνε πώ λειτουργεί το σύστημα. Μπήκαν σε αυτόν τον απόκριφο λεγόμενο κήπο τη συμμετοχή τη εγγραφή στι εκλογικέ λίστε. Το να κατηγορούνται γυναίκες για την ε, μη εκπροσώπησή τους είναι λάθος. Άκουσα τέτοιε κατηγορίε και στη Μάλτα και στο Μαρόκο και στη Γαλλία ακόμη είναι δεκτυπώνονται ει βάρο των γυναικών. Δεν, φτάνει δεν φταίνουν οι γυναίκε αν δεν υπάρχουν αρκετέ γυναίκε υποψήφοι. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Γάλλος, ο άνδρας, συγγνώμη, ψηφοφόρος δεν ψηφίζει για γυναίκα ψηφοφόρο. Βέβαια ούτε για άντρα ψηφοφόρο ψηφίζει, δεν θα ψηφίσει με βάση το φύλλο, θα ψηφίσει γιατί είναι επιχειρηματία ο υποψήφιο, θα ψηφίσει γιατί είναι γεωργό, γιατί είναι εκπρόσωπο του Δίνα ή του τάδε κλάδου. Αλλά η γυναίκα θα ψηφίσει και την γυναίκα, με το κριτήριο δηλαδή του φίλου. Η δράση λοιπόν, η ώρα για δράση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια προσπάθεια να εξεταστούν τα ποσοστά επιτυχίας των γυναικών στις ευρωεκλογές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν άντρες ή γυναίκες ανάλογα με την ε, λίστα ή την εκλογική περιφέρεια στην οποία κατα... Ε, ε, εγγράφονται υποψήφοι. Για να εκλεγούν 5% γυναίκες σε μια βουλή χρειάζονταν 63% γυναίκες υποψήφοι σε έναν εκλογικό κατάλογο για να βγει αποτέλεσμα 5% τουλάχιστον εκλεγωμένων για να καταλάβετε αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, όταν αρχίσουν οι γυναίκε να πλησιάσουν το 50%, αρχίζει ο κόσμο και φοβάται. Και γυναίκε ακόμη αισθάνονται ανησυχία, γιατί ανεβαίνουν τα ποσοστά των γυναικών. Εγώ, προερχόμενη από σκανδιναβική χώρα, ακόμη με τα δικά μα τα δεδομένα, πάλι διαπιστώνω ότι ο κόσμο φοβάται και αισθάνεται ανησυχία όταν οι γυναίκε ανεβαίνουν, ε, ανεβάζουν την παρουσία του στην πολιτική ζωή, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Όταν έχουμε μια πολιτική επιτροπή, ένα κοινοβούλιο κτλ. με 30-35% συμμετοχή των γυναικών, και 65 ως εκ τούτου ανδρών, πολλοί είναι αυτοί που θα πούνε «Α, εντάξει, ισότιμη συμμετοχή, πολύ καλά». Αν όμως αντίστροφα είναι 65% οι γυναίκες και 35% οι άντρες, α, θα πούνε «Αυτό είναι γυναικοκρατία». Και προφανώς κακό πράγμα. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, δούμε το σύστημα αυτό του, ε, της εγγραφής στην εκλογική λίστα, πώς λειτουργεί αυτός ο μυστικός κήπος τον οποίο προαναφέρθηκα, που σημαίνει τελικά ότι για να μπει μια γυναίκα σε έναν εκλογικό κατάλογο και να έχει την ελπίδα να εκλεγεί σε μια εκλογική αναμέτρηση, πρέπει να έχει ξεκινήσει την εκστρατεία της και τον αγώνα της δύο χρόνια πριν, δηλαδή να έχει μπορέσει να πείσει αυτούς που πρέπει να πείσει για να την ε, βάλουν υποψήφια στην λίστα. Μετά επίσης, κοιτάξτε λίγο, ε, όταν γίνονται στο Συμβούλιο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλε συναντήσει ή όταν παίρνουν τη μεγάλη φωτογραφία, τη λεγόμενη οικογενειακή με όλου του αρχηγού παδών και κυβέρνησεων. Πόσε είναι οι γυναίκε που θα δείτε εκεί πάνω στη φωτογραφία. Ή σε επίπεδο κοινοβουλευτική επιτροπή, με 4.000 υποεπιτροπέ που διαθέτει και που εργάζονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχουν καν στατιστικέ επαρκεί που να μπορέσουμε να μελετήσουμε για να δούμε τι ε, εκπροσώπηση έχουν οι γυναίκες και οι άντρες στα όργανα αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμως ε, από τα στοιχεία που μπορέσαμε να συλλέξουμε βλέπουμε ότι η ισότιμη μεταχείριση των φύλων ή η συμμετοχή μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς και πολλαπλούς ε, όρους και μορφές και το χειρότερο που θα μπορούσε κανείς να κάνει θα ήταν να επιβάλλει ένα σύστημα ποσοστώσεων φύλων που δεν θα ήταν σύμφωνο με το εκλογικό σύστημα, γιατί αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα και ενοχλήσεις ε, στους πάντες. Τελικά θα έκανε περισσότερη ζημιά δηλαδή. Μέχρι στιγμή λοιπόν οι ποσοστώσει υπέρ των φύλων υπάρχουν σε αρκετέ χώρε, σε πέντε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τις ε, λεγόμενες εθελούσες ποσοστώσεις, ε, μη εθελούσες ποσοστώσεις και απουσία ποσοστώσεων, ανάλογα με τη χώρα και με το κόμμα. Υπάρχουν τρία μόνο κόμματα στην Ευρώπη που έχουν εθελούσιο σύστημα ποσοστώσεων και 16 που έχουν μη εθελούσιο. Πιστεύω λοιπόν ότι το σύστημα των ποσοστώσεων για τα φύλλα πάντα ε, έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό πρώτον διακρίσεις βάρος των ανδρών. Και ακούω να ξεκινούν ορισμένοι να φωνασκούν ναι, για ένα λεπτό όμω, σα εξηγήσω. Εδώ στο, στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, το οποίο προέρχεται το παράδειγμα μου, έχουν, έχουμε ένα σύστημα ισορροπημένο 50% άνδρε, 50% γυναίκε. Όσοι άνδρε, τόσε γυναίκε. Και δεν υπάρχει τρόπος ε, να περάσει κανείς πιο πάνω ή πιο κάτω στη λίστα. Δεν είναι θέμα δηλαδή θέσεως στην εκλογική λίστα. Πάντοτε ό,τι και να γίνεται θα εκλέγεται ένας άντρας και, και μία γυναίκα αντίστοιχα. Το σύστημα όμω αυτό τη ποσόσταση, όσο ισότιμη και να είναι η συμμετοχή των ε, φίλων, δεν εξασφαλίζει ε, νομιμοποίηση των αποφάσεων που θα λαμβάνονται, γιατί οι αποφάσει μπορούν να ληφθούν ε, και να είναι κακέ ή καλές. Υπάρχουν διαφορετικά παραδείγματα λοιπόν ή υποδείγματα ποσοστώσεων σε διάφορε χώρε η Γαλλία ήταν ένα κακό, καλό σύστημα. Με, είχε απογοητεύσει στην αρχή με το 8% στην αρχή και το 12% στη συνέχεια των εκλεγωμένων γυναικών που δεν αντιστοιχούσαν φυσικά στην ε, ε, διαδικασία που θα έπρεπε να έχει εισαχθεί. και στο Ηνωμένο Βασίλειο ιδιαίτερα όπου έχουμε το σύστημα της μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας ε, υπάρχει τεράστια δυσκολία να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών γιατί βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε σύστημα ποσοστώσεων σε μονοεδρικά συστήματα. Η Ισπανία επίση, η οποία τώρα έχει καταπληκτικά αποτελέσματα να επιδείξει και έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα τη ισότητα, ανδρών και γυναικών με άλματα μεγάλα στην ιστορία που δεν γνωρίσαμε ούτε εμεί στις χώρες ε, του αρκτικού κύκλου. Πλην όμως τα αποτελέσματα του συστήματο των ποσοστώσεων τη Ισπανίας ήταν 36% ε, ε, εκλεγόμενες γυναίκε στο παρελθόν και 36,3% μετά την εισαγωγή του συστήματο των ποσοστώσεων. Άρα λοιπόν όλο αυτό το σπουδαίο σύστημα που έλεγε ότι, ότι από τους πρώτους πέντε τουλάχιστον δύο θα πρέπει να είναι γυναίκες και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί σε τελευταία ανάλυση μην ξεχνάμε ότι κάποια κόμματα δεν εκλέγουν πάνω από δύο ή τρεις υποψηφίους τους ε, στο κοινοβούλιο και άρα από αυτούς τους δύο ή τρεις, το πολύ δύο να είναι γυναίκες, δεν άλλαξε άρδερ το πολιτικό πεδίο. Άρα υπογραμμίζω ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό σύστημα ποσοστώσεων και δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί η επιτυχία στους αγώνες αυτούς ε, η εισαγωγή ενό οποιοδήποτε συστήματο ποσοστώσεων. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα ποσοστώσεων. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει κανεί με την διάγνωση των προβλημάτων. Γιατί υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι υπάρχουν νέε αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις οποίες ε, παρουσίασε και η Μάρκοτ Βάλστρομ ε, πρώτη από όλους και μπορούμε να αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνεια για τις προσπάθειές της. Γιατί γιατί όταν μιλούν μεταξύ τους άνδρες πολιτικοί για να ορίσουν ε, εκλογικό κατάλογο, για άνδρες υποψηφίους θα συζητήσουν, όχι για γυναίκες. Δεν θα έχουν μέλημα τη γυναίκα ή το ρόλο της. Γι' αυτό λοιπόν όταν μπει κανείς σε αυτό το μυστικό κύκλο των ληστών, τα προβλήματα είναι πολλά πρέπει να, υπάρχουν ε, πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση όχι μόνο με βάση το φύλλο, αλλά και με βάση τη δραστηριοποίηση σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Πρέπει να έχουμε και από τα εκλογικά συνδικάτα, πρέπει να έχουμε και από τη γεωργία, πρέπει να έχουμε και από το χώρο τη μηχανία εκπροσώπηση. Και αυτό και για το ένα φύλλο και για το άλλο. Και αυτό ε, σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται υποτίθεται είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, βαθμός δεξιοτήτων των γυναικών για να μπουν σε τέτοιου είδους θέσεις. Όμως αυτό δεν ευσταθεί γιατί οι γυναίκες στην Ευρώπη έχουν δεξιότητες προσόντα, ικανότητες ισότιμα με αυτά των ανδρών και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να υποεκπροσωπούνται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η ε, καταγραφή, η θέση στον ε, κατάλογο τον εκλογικό. Αλλά μην κατηγορείτε τις γυναίκες όταν δεν επιτυγχάνουν. Μην ορίσετε στην τελευταία ανάλυση κάποιο συγκεκριμένο άντρα όταν δεν εξασφαλίζεται η ισότιμη ε, μεταχείριση. Όχι, αλλάξτε τους θεσμούς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Και εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφαση. Πολλά αλλάζουν στον κόσμο. Και σας είπα νωρίτερα ότι η Ευρώπη δεν είναι πρώτο πόρος στα θέματα των γυναικών, αλλά με χαρά βλέπω ότι τουλάχιστον και στην Ευρώπη σημειώνεται πρόοδος. Χωρίς βέβαια να ισχυρίζομαι ότι οι ποσοστώσεις είναι οι πανάκια ή ότι μπορεί να επιλύσουν κάθε πρόβλημα. Όμως πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα και να διαρωτούμεθα γιατί υπάρχει υποεκπροσώπηση των γυναικών. Μια σωστή διάγνωση μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σωστή αντιμετώπιση. Και να περάσετε πολύ καλά την 8η Μαρτίου όλες σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία καθηγήτρια Ντάλερουπ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. πήγε έμπνευση από αποτέλεσε για τις ευρωεκλογέ στις οποίες αποδιόμαστε τώρα στις χώρες μας και στο δεύτερο τμήμα των ε, συζητήσεών μας θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία και σε εσάς πάλι να μιλήσετε αγαπητοί και αγαπητές προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες μην ξεπερνώντας όμως τα δύο λεπτά και θα κάνουμε την αναλλαγή που συνηθίζουμε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων ή ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρώτα και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Γενικών και ε, Ίσων Ευκαιριών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή. Ακούσαμε τι γίνεται με την επιρροή των γυναικών στα κράτη-μέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Αυτό που ανησυχεί είναι η σχνήση προσώπηση γυναικών ιδιαίτερα στις ευρωεκλογές. Λίγες γυναίκες ε, επίση ψηφίζονται. Γι' αυτό το 55% θα πρέπει να δουλέψουμε, θα πρέπει να επιδείξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά γυναικεία δικαιώματα. Θα πρέπει στα κρατη μας και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δείξουμε ότι σήμονται βήματα σχετικά πούμε με τις μισθούς, τις αμοιβέ, με την απασχόληση γυναικών, το ποσοστό τους. Γιατί θα πρέπει να τους δείξουμε ότι εργαζόμαστε και για τα ηλικιωμένα άτομα, για τη σεξουαλική ε, για την σκλαβιά λόγω του φύλου. Θέλουμε να δείξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη βελτίωση ποιότητα, τη ζωή των γυναικών. Όλα αυτά που γίνονται γιατί βλέπουμε ότι οι άνδρε αποφασίζουν και κατασκευάζουν για άνδρε. Ε, να σα πω και μένα επίκαιρα πράγματα να μιλάμε για την κρίση, α πούμε, την οικονομική. Εγώ συναντήθηκα με μια ομάδα εμπειρογνωμών της Επιτροπής για να δούμε το θέμα της απλής της κρίσης και αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελείται από οκτώ άνδρες, άνδρες μόνο. Για τη λύση λοιπόν της κρίσης τι γίνεται, οι άνδρες θα αποφασίσουν, οι άνδρες θα προχωρήσουν, οι άνδρες που είναι ακόμα και για την ε, θέματα εκμετάλλευσης ε, το ένα το άλλο και θα πρέπει να έχουμε πραγματογνωμοσύνες και από πλευράς γυναικών, πώς βλέπουν εκείνες την κατάσταση και τι προτείνουν για τη λύση και να δούμε και για τα θετικά σημεία, τουλάχιστον στο κόμμα μου της αριστερά στη Σουηδία, γνωρίζουμε ότι οι εκλογείς μας άνδρες και γυναίκες απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες σε ε, υψηλές θέσεις και τα ψηφοδέλτιά μας εκεί κυριαρχούν και οι γυναίκες γιατί το απαιτούν οι εκλογείς. Χρειάζεται μια καλύτερη ισορροπία για όλα τα κόμματα βέβαια. Θα πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό το έργο αυτό, να επιτευχθεί σε όλα τα κράτη-μέλη και τα δικαιώματα των γυναικών να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να σπάσουμε αυτήν την λυσίδα διαθρωτικής διάκρισης ε, λόγω φύλου με υψηλών και υποφέρουν οι γυναίκες από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορεί να λάβει το λόγο εκπρόσωπος του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου, κ. Πολ Χέρνιεφ, μέλος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να μιλήσω για τις ελπίδες που έχω με τρόπο έτσι πολύ άνετο, φιλικό και ανεπίσημο. Όλα αυτά που άκουσα πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα. είναι σημαντικό να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε σε πραγματικά ίσα δικαιώματα που απολάβουν τελικά οι γυναίκες και οι άντρες. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στα θέματα που έθεσαν η κυρία Σβένσον και η καθηγήτρια από την ε, Σουηδία. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία. Στα, στις τελευταίες εκλογές στις οποίες συμμετείχε το κόμμα μου, το οποίο δεν είναι ούτε κεντρό ούτε αριστερό, αντιμετώπισε ένα αρκετά ιδιάζον φαινόμενο. Σε μία εκλογική περιφέρεια, μία νεαρή κυρία, αρκετά ευηδής, ήταν υποψήφια και αυτό μας εξασφάλισε την πρώτη θέση σε αυτή την εκλογική περιφέρεια σκεφτήκαμε ότι τα γυναικεία πρόσωπα ε, δρούν ως ε, απίστευτος καταλήτης για τους ε, εκλογείς, τους πρόχνουν στο να προσφύγουν στις, να προσφύγουν στις κάλπες. Ένα γυναικείο χαμογελαστό πρόσωπο είναι πραγματικά πολύ πιο ελκυστικό από τα συνοφιωμένα αντρικά πρόσωπα. Ζητώ συγγνώμη που σας μιλάω για αυτά τα πράγματα. Ε, σας μιλάω για ένα κόμμα, για ένα δεξιό κόμμα. Αυτό λοιπόν, ε, αυτή η εμπειρία μας έκανε να σκεφτούμε ότι πρέπει να βάλουμε επικεφαλής του καταλόγου μας μια γυναίκα, γιατί πραγματικά η γυναίκα θα μας εξασφαλίσει την νίκη. Οι γυναίκες ε, θα μας βοηθήσουν. Είμαι πεπισμένος ότι οι γυναίκες υποψήφιες στις εκλογές εκφράζουν πολύ, πολύ πιο καθαρά το πολιτικό μήνυμα που θα θέλαμε να περάσουμε. Είμαι πεπισμένο βαθιά για αυτά που σας λέω. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε τόσο πολύ την απουσία των ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις θα λειτουργήσουν ούτως ή άλλως στο βαθμό που οι γυναίκες λειτουργούν καλά και δουλεύουν καλά. Σα ευχαριστώ. Τον εκπρόσωπο του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικέ φορέ έχουμε την εντύπωση ότι λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Εν γέννη, όταν έχουμε τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας, συζητούμε ποια είναι η θέση τη γυναίκα και σαν να παίζουμε συνέχεια, σαν να έχει χαλάσει ταινία και να γυρίζει γύρω-γύρω να ακούμε τα ίδια πράγματα. Έτσι λοιπόν, Ίσως θα έπρεπε να στρεφούμε περισσότερο στις βάσεις, τους λόγους για την μη ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Οι λόγοι είναι όχι μόνο η νομοθεσία. Λόγος είναι πέραν της νομοθεσίας η στάση μας και στο Εθνικό ή στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο όταν έρχεται η ώρα της εκλογής. Και αυτά είναι προβλήματα τα οποία με την ε, λύση του gender mainstream μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε γιατί θεωρούμε ότι ε, η νομοθεσία μπορεί μεν να ορίζει από το 59 στην πατρίδα μου ότι δεν μπορεί να υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών αλλά τα αποτελέσματα, τα ουσιαστικά αποτελέσματα στην εκπροσώπησή μας δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά. Και οι τάσεις μπορεί μεν να είναι υπέρ των γυναικών, από καιρού εις καιρών όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και οπισθοδρομήσεις. Βέβαια δεν είναι η νομοθεσία πάντοτε το... Ε, ο τρόπος ή η πανάκια να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα. Ένα από τα, ένα, μία από τις λύσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε θα ήταν το σύστημα των ποσοστώσεων όπου βλέπω πως χρειάζεται να έχουμε πάντα υπόψη ότι ο δρόμος από την γιούρα, ε, ισότιμη μεταχείριση έως την de facto ισότιμη μεταχείριση, ο δρόμος είναι μακρύς. Και η ευθύνη μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή τα εθνικά είναι βεβαίως πολύ μεγάλη η ευθύνη που έχουμε αναλάβει από εμά μόνο θα προχωρήσει, μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα και δεν μπορεί κανείς άλλος να κάνει τη δουλειά για μας, στη θέση μας. Γιατί όσο καλή και αν είναι η νομοθεσία, όσο ουσιαστική και ε, ισότιμη νομοθεσία δεν ε, φέρνει κανένα αποτέλεσμα εάν δεν εφαρμόζεται. Σωστά. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ και τώρα η κυρία Φανσουάς Καλτρών από το Γαλλικό Κοινοβούλιο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την συνάντηση που επέτρεψαν σε όλους μας να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας μιλήσω για την θεώρηση της Γαλλίας, για τους νόμους που έχουμε στη Γαλλία ε, και να σα απαντήσω στα ερωτηματικά που θέσατε. Καταρχάς ξεκινήσαμε από τη διαπίστωση ότι σε ό,τι αφορά τη θέση της γυναίκας και την δίκαιη εκπροσώπηση της γυναίκας στην πολιτική, δεν θα μπορούσαν να εξελιχθούν φυσιολογικά, ιστορικά. Είδαμε ότι μέσα σε 50 χρόνια δεν κερδίσαμε καθόλου νέες θέσεις και επομένως ότι θα πρέπει να λάβουμε μέτρα, κίνητρα Γι' αυτό ακριβώς ο νόμος για την ισότητα ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε σε, όλους, σε όλες τις εκλογικές μάχες που δίνονται με κατάλογο. Νομίζω ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, ε, δεν τάραξε τις νοοτροπίες, γιατί ε, η κοινωνία μας είναι έτοιμη. Οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες είναι έτοιμοι να ψηφίσουν για γυναίκες. Εκεί που υπήρχαν περισσότερα προβλήματα ήταν σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων. Υπάρχει μάλιστα ένα δεύτερο μέτρο ε, που πήρε το Σοσιαλιστικό Κόμμα στο οποίο ανήκει, ανήκω για όλες τις ονομαστικές ψηφοφορίες και κυρίως ε, για τις ε, βουλευτικές εκλογές. Ένα μέτρο λοιπόν να κρατήσουμε κάποιες εκλογικές περιφέρειες για γυναίκες. Εκεί οι γυναίκες, οι άντρες δεν θα μπορούσαν να είναι καταρχήν υποψήφοι. Αυτό έβαλε κάποια, έθεσε κάποια ερωτηματικά. Δύο εκλογές οργανώθηκαν έτσι. Ε, σε, στο 50% των εκλογικών περιφερειών λοιπόν κατεβήκαν οι γυναίκες σε όλη τη γαλλική επικράτεια. Εκλέχτηκαν αυτές οι γυναίκες. Μερικές φορές οι εκλογικές ε, περιφέρειες θεωρούνταν δύσκολες και λέγαμε ας πούμε αποκλείεται να εκλεγεί γυναίκα σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Και όμως εμείς αποδείξαμε ότι γίνεται. Σήμερα λοιπόν οι γυναίκες απέδειξαν ότι δεν υπάρχουν ταμπού, μπορούν να εκλεγούν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας μας και όμως δεν υπάρχουν ταμπού γιατί οι εκλογείς, άντρες και γυναίκες αναγνωρίζουν τα πρόσφατα των γυναικών. Και για όλα αυτά τι θα ήθελα να πω, μπράβο, ζήτω οι γυναίκες. Ε, Ευχαριστώ πολύ και τώρα νομίζω μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Γκρόινερ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, χρόνια πολλά ήμουν παρούσα σε διεθνείς ημέρες της γυναίκας και αντίστοιχες ε, <clears throat> και αντίστοιχε εκδηλώσει. Αντίθετα όμω από την κυρία Λούλινγκ, έχω μένει πάντοτε στο ίδιο κόμμα, στην ίδια πολιτική ομάδα, τη Σοσιαλιστική. Για την ε, <clears throat> Επιτροπή των δικαιωμάτων των γυναικών, ε, ξέρουμε ποιοι είναι οι αγώνες μας, ξέρουμε πόσο ακόμα δρόμο έχουμε να διανύσουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στην αμοιβή που παίρνει μια γυναίκα ή ένας άντρας για την ίδια δουλειά, ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν στην εκπροσώπηση, στις ευρωεκλογές, στις εθνικές εκλογές, σε πολλά θέματα βέβαια η κατάσταση πάει προς το χειρότερο. Με αυτά που ακούμε μερικές φορές και από υπουργού διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να επιληθούν μόνο με ευχολόγια. Είδαμε και τον Τσέχο Υπουργό εδώ πέρα. Δυστυχώ δεν ε, είναι πια εδώ για να συζητήσουμε μαζί του. Σε μερικέ ημέρε που συνεδρία το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων να δούμε τι θα προσφέρει αυτό η λυπή Υπουργή για τα θέματα τη γυναίκα, Αλλά πάντως στόχοι τη της Λισαβόνας δεν θα επιτευχθούν εάν δεν υπάρχει ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Εγώ εκπροσωπώ τη Γερμανία αν και βλέπω ότι δυστυχώ το Γερμανικό Κοινοβούλιο δεν έχει εκπρόσωπο εδώ σήμερα. Είναι κενά τα έδρανα που έχουν για τις για τους Γερμανούς και τις Γερμανίδες ε, εθνικούς βουλευτές. Η κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα, η οικονομική κρίση, θα ήθελα να σημειώσω όμως, φαίνεται ότι έχει προκληθεί από υπερβολικό βαθμό τεστοστερώνης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ίσως θα έπρεπε να δούμε εκεί ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης για την οικονομική κρίση σε όποιες χώρες επιτοπλίστων του Βόρειου Αρκτικού Κύκλου υπήρχαν γυναίκες σε ηγετικές θέσεις δεν είχαμε τόσο σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν είχαμε καταρρεύσεις οικονομιών ή ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το ίδιο πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένα και καλά μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές διακρίσεις βάρος των γυναικών. το κριτήριο της ισότιμης μεταχείρισης των ε, Τη μάλλον τη θετική διάκρισης των γυναικών δεν το έχει κάνει δεκτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει έννοια των διακρίσεων ε, γενικά, αλλά όχι ιδιαίτερα στον χώρο εργασία. Αυτό δεν έχει αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ε, ε, και αν δεν αναγνωριστούν ε, οι διακρίσει που πράγματι υφίστανται ει βάρο των γυναικών στον χώρο εργασία, πώ είναι δυνατόν να τι αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω ότι θα είναι περισσότερε οι γυναίκε οι οποίε θα μπορέσουν να προχωρήσουν στον αγώνα αυτόν για να έχουμε περισσότερη ε, ε, πρόοδο. Ελπίζω δηλαδή να έχουμε και περισσότερε ε, γυναίκες ευρωβουλευτέ μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Αλλά πάντως πρέπει να σημειώσω ότι χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά για να κερδίσουμε στον αγώνα αυτό. Εάν δούμε πόσο γρήγορα διατέθηκαν τα δισεκατομμύρια που παρένα να καλύψουν τις τα προβλήματα, εν περιπτώσει, ή τις ελλείψεις που προκάλεσαν άντρες επικεφαλής ε, μεγάλων οργανισμών, ομίλων και εταιριών, ε, και με πόση βραδύτητα προχωράει το θέμα των γυναικών, αγανακτούμε πραγματικά, τουλάχιστον εγώ αγανακτώ πραγματικά. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε και σε επίπεδο ανδρών αυτούς οι οποίοι θα λαμβάνουν αποφάσεις με προσανατολισμό το φύλλο που θα έχουν μια ευαισθησία δηλαδή απέναντι στις γυναίκες όχι γιατί εξορισμού η γυναίκα πρέπει να είναι καλύτερη αλλά γιατί πρέπει να έχει εξίσου καλές ευκαιρίες να προχωρήσει αν έχει τις ίδιε τις ίδιες ικανότητες έτσι ώστε να προχωρήσουμε χέρι με χέρι και ισότιμα για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρένερ. Η εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρακαλώ. Η κυρία Αράπαγλου μπορεί να λάβει το μικρόφωνο. Είναι μέλος της μόνιμης Επιτροπής για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των νέων. Πριν όμως, πριν όμως του δώσω το λόγο στην κυρία Βουλευτή, θα ήθελα, πριν όμω δώσω το λόγο στην κυρία Αράπογλου, θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μόλι ήρθε μέσα στην Ολομέλεια και βέβαια μέλο τη Επιτροπή μα των Δικαιωμάτων των Γυναικών και των Ίσων των Φίλων, την κυρία Κράτσα. Καλώ ήρθατε και χαιρόμαστε πολύ που σα βλέπουμε εδώ. Κυρία Αράπογλου, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε και να δώσω το λόγο στην κυρία Αράπογλου. Είμαι η μοναδική κοφή βουλευτής ε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου και η τέταρτη στον κόσμο. Και φυσικά θα ζητήσω λίγο την κατανόησή σας λόγω της χρήσης νοηματικής ε, ως προς το χρόνο. Έχω κλείσει ήδη δύο χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν, δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι μεγάλη τιμή για την ε, είναι μεγάλη τιμή για την γιορτή της γυναίκας, τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας που οργανώνεται μια τέτοια εκδήλωση. Οι διεκδικήσεις των γυναικών για τα δικαιώματά τους μετράνε πάρα πολλά χρόνια. Η γυναίκα έχει καθιερωθεί ιστορικά μέχρι σήμερα ως μια, ένα άτομο που συνεχώς παλεύει για τα δικαιώματά του και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις προτεραιότητες και τις συνθήκες ζωής τους ο ρόλος της γυναίκας στη ζωή μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί η γυναίκα έχει και πολλαπλούς ρόλους. Είναι σύζυγος, μητέρα, εργαζόμενη. Και φυσικά η γυναίκα έχει πολύ μεγάλες ευθύνες μέσα στην ε, κοινωνική ζωή. Πρέπει να φροντίζει για την ανατροφή των παιδιών, και έχει πολλούς ρόλους όπως είπα. Γι' αυτό και οι άντρες αντίστοιχα πρέπει να εκτιμούν αυτή την πολλαπλή συμβολή των γυναικών στην ε, ζωή και να ε, βλέπουν και τις ανάγκες τους. Πιστεύω ότι ε, στις ε, επερχόμενες ε, ευρωεκλογέ θα πρέπει η συμμετοχή των γυναικών να είναι μεγαλύτερη και να αναγνωριστούν τα δικαιώματα, των γυναικών να, να θέτουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται και να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική ζωή. θα πρέπει να τη δίνονται, τα δικαιώματα να μπορεί να συμμετέχει και στην πολιτική ζωή και στην οικογενειακή αλλά και στην καριέρα. Και φυσικά, όπως ξέρετε, στην ελλάδα προσπαθούμε πάρα πολύ και παλεύουμε για τα δικαιώματα των γυναικών και για τη συμμετοχή τους και μέσω του αναπηρικού κινήματος. Στην Ελλάδα, μέσω, της, του μέσω του τετραετούς ε, προγράμματος για την προτεραιότητα μέσα μέσω του τετραετού προγράμματο εθνικέ προτεραιότητε, πολιτική και Άξονες Δράσης για την Ισότητα των Δύο Φύλων 2004-2008 προσπαθήσαμε και κερδίσαμε πολλά ε, πράγματα, ειδικότερα για τις ε, γυναίκες ε, που είναι άτομα με αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή. Για παράδειγμα, γυναίκες που φροντίζουν άτομα με αναπηρία ενήλικα τέκνα να μπορούν να δηλώσουν ω έδρα την οικία του είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τι διακρίσει, και αυτέ οι διακρίσει πρέπει να σταματήσουν. Επίση, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε και να σταματήσει είναι η βία κατά των γυναικών. Και είναι σημαντικό από όλε τι χώρε, και αυτό με ενδιαφέρει πραγματικά, είναι να δούμε η κάθε χώρα τι θέσει εκπροσωπεί, ποιος, είναι η στόχη της, ποιοι είναι οι στόχοι της κάθε χώρας, τι προτείνει συγκεκριμένα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μας για ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών. τι θα συμβουλεύαμε μια γυναίκα που θέλει να είναι ενεργή στην ε, επαγγελματική της ζωή, να έχει την καριέρα, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσει και τους ρόλους τους υπόλοιπους που έχει. Τι θα συμβουλεύαμε, ποιε είναι οι πολιτικές της κάθε χώρας για τη γυναίκα. Ποια είναι η θέση της κάθε χώρας. Θα, θα ήθελα να το ακούσω πολύ συγκεκριμένα. Και τις απόψεις της κάθε χώρας. Και τις απόψεις του, της κάθε πολιτικού. Για μένα αυτό είναι σημαντικό, να ακούμε συγκεκριμένα πράγματα γιατί εδώ μιλάμε για τις γυναίκες που παλεύουν και δεν είναι όπως αντίστοιχα ένα άντρα που έχει λιγότερες υποχρεώσεις. Οι γυναίκες έχουν περισσότερες υποχρεώσεις. Οι, οι άντρες σκέφτονται με το αριστερό ε, μέρος του τους. Οι γυναίκες με το δεξί. Αυτό τι σημαίνει. Πρέπει να κάνουμε διαχωρισμούς. Ποιος έχει τον δυναμισμό, ποιος είναι πιο αποφασιστικός. Τη δύναμη την έχει η γυναίκα τη γυναίκα γιατί παίζει πάρα πολλούς ρόλους στη ζωή και γι' αυτό ξέρει πώς να παλεύει. Ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ε, Θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ράπογλου για όσα μας είπε. Η κυρία Ράπογλου συμμετείχε στην ε, συνάντησή μας και πέρυσι χαιρόμαστε που και φέτος είναι παρούσα. Η κυρία Κράτσα το έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και εγώ σήμερα μαζί σας σε αυτή την εκδήλωση που έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί γίνεται λίγες μέρες πρώτης Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας που μας καλεί σε απολογισμούς, προβληματισμούς, σκέψεις, προγραμματισμούς αλλά και γίνεται και λίγους μήνες πρώτων ευρωεκλογών. Γι' αυτό το θέμα μας είναι επικεντρωμένο και γι' αυτό η συνάντησή μας έχει μεγάλη σημασία διότι πρέπει να ανταλλάξουμε σκέψεις και προγραμματισμό να συμβάλλουμε ούτως ώστε στις ευρωεκλογές να αναδειχθούν περισσότερες γυναίκες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να διεκδικήσουμε οι γυναίκες αυτές να παίξουν σημαντικούς ρόλους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αυτό συνήθως γίνεται από επιλογές κομματικές και επιλογές των αντιπροσωπιών τους, δεν ανταποκρίνεται πάντα στις δικές τους επιδιώξεις και στη δική τους αξία Οπότε η δέσμευση των πολιτικών κομμάτων για το ρόλο που θα παίξουν οι αντιπροσωπείες τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να κάνει και με τη θέση που τα κόμματα δίνουν στις γυναίκες. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε και πιστεύω ότι για να εξετάσουμε την κατάσταση σε κάθε χώρα μέλος όπως μόλις είπε η κυρία Ράπογλου πρέπει να συνεργαστούμε με βάση κάποια δεδομένα, τα στατιστικά στοιχεία, της μελέτης, την ανταλλαγή πληροφοριών που θα έχουμε και πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το ευρωβαρόμετρο το οποίο ειδικά ε, πραγματοποιήθηκε ειδική έρευνα για τις ευρωεκλογέ και την δημογραφική και κοινωνιολογική μελέτη την οποία έχουν κάνει οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου το δώσαμε χθε στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε σήμερα γιατί οι υποχρεώσει μου δεν μου επέτρεψαν να είμαι από την αρχή αυτή τη εκδήλωση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το δούμε στη βάση του και στο πλαίσιο κάθε, κάθε χώρα. Η μελέτη αυτών των στοιχείων, οι, οι σκέψει, τα συμπεράσματα που θα συλλέξουμε είναι σημαντικά για την προεκλογικό μα αγώνα, διότι εκεί θα δούμε ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται πάνω απ' όλα για συγκεκριμένα θέματα, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής τους και την καθημερινότητα της οικογένειας, όπως η ανεργία, η αγοραστική δύναμη, η κοινή επιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διαζευμένων ζευγαριών και θα δούμε επίσης ότι άνδρες και γυναίκες αναγνωρίζουν ότι η κοινωνία μας είναι ανδροκρατούμενη. 86% των γυναικών 76 των ανδρών το αναγνωρίζουν. Και το 50% των γυναικών κάνουν έκκληση για μια ισόρροπη συμμετοχή, όχι μόνο για να δικαιωθούν οι αγώνες τους, αλλά γιατί πιστεύουν ότι η κοινωνία θα γίνει καλύτερη. Αυτά είναι θέματα τα οποία εμεί έχουμε ξανασυζητήσει μεταξύ μα. Είμαι σίγουρη ότι μοιραζόμαστε τι σκέψει και τι διαπιστώσει αυτέ. Έχει σημασία να τι δούμε στην εθνική πραγματικότητα και να τι αξιοποιήσουμε για τι ευρωεκλογέ. Η περίοδο λοιπόν που έρχεται είναι μια περίοδο και δράση και δεσμεύσεων για όλε μα και πρέπει αυτά να τα μεταφέρουμε στα πολιτικά μα κόμματα, στην κοινωνία μα και έτσι θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Περισσότερες γυναίκες, περισσότερη θέση στο διάλογο, στη συζήτηση και στις δεσμεύσεις για θέματα που αφορούν τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ε, συνεργασία θέλετε σε επίπεδο ευρωπαϊκό ή σε κάποια χώρα μέλος που ήδη ετοιμάζει την προεκλογική της καμπάνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, την κυρία Κράτσα. Τώρα δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Είναι μέλος της Επιτροπής Γυναικών και των Δικαιωμάτων Γυναικών. Η κυρία Κουτό, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή τη συνεδρίαση. Θα, θα προσπαθήσω να θέσω δύο ερωτήματα στη συζήτησή μα. Πώ θα κινητοποιήσουμε τα πολιτικά κόμματα και πώ θα κινητοποιήσουμε τι γυναίκε να ασχοληθούν με την ε, πολιτική. Πώ θα κινητοποιήσουμε τα κόμματα με τον νόμο. Ε, με το γαλλικό σύστημα σύνταγμα ε, δεν επιτρέπονται οι ποσοστώσεις. Εμεί ψηφίσαμε την ισότητα. Και νομίζω ότι είναι καλό αυτό, γιατί οι ποσοστώσεις είναι, είναι ένα εργαλείο για να καταπολεμήσουμε τις ε, διακρίσεις, αλλά η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι μια μάχη που πρέπει να δίνεται σε όλα τα επίπεδα. Πώς θα κινητοποιήσουμε τα πολιτικά κόμματα, υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ε, καταρχάς, ε, με πρόστιμα. Το εφαρμόσαμε στη Γαλλία. Τα κόμματα ε, πληρώνουν πρόστιμα όταν υπάρχουν αρκετέ υποψήφιε. Και δεύτερο, ε, η μη σώρευση των αξιωμάτων. Ε, στη διάρκεια του χρόνου και ε, διαδοχικά εκλογικά αξιώματα δεν υπάρχει δυνατότητα να τα συσσωρεύσει κανείς. Επομένως έτσι απελευθερώνται θέσεις για νέες ε, για γυναίκες, για νέες πολιτικούς. Δεύτερον, πώς θα κινητοποιήσουμε τις γυναίκες να ασκήσουν πολιτική. Δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται κατά ανάγκη από μόνες τους για την πολιτική. Εδώ νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ε, στο βοηθώντας τις γυναίκες να ασκήσουν τα αγωνικά τους δικαιώματα. Θα πρέπει οι γυναίκες ε, απελευθερωνόμενες και αποκτώντας περισσότερο χρόνο επειδή τα καθήκοντα θα τα μοιράζονται με τους άντρες να βοηθηθούν για να ασχοληθούν με την πολιτική. Πρόεδρος. Η κυρία Εστρέγια, η αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ένα χρόνο μετά να που και πάλι συζητάμε για τα ίδια θέματα και επαναλαμβάνουμε τα ίδια επιχειρήματα. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία να έχουν επηρεάσει θετικά την κατάσταση για ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για τα υπόλοιπα, όταν άκουσα να μιλάει πρόσωπος από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο, αυτό μου κάνει ακόμα πιο σίγουρο την άποψή μου ότι χρειάζεται πλατύτερη συζήτηση για να δώσουμε τη μάχη μας κατά των ε, παλαιοληθικών εκφράσεων. Ε, τα ίδια δικαιώματα έχουν οι γυναίκες όπως και οι άνδρες για να πετύχουν στη σταδιοδρομία τους, να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων και στην πολιτική ζωή και στην οικονομική ζωή. Και όχι μόνο και μόνο ε, να ομορφαίνουν τα ψηφοδέλτια. Δεν είναι καλυστία οι εκλογές. Είναι μια απόδειξη αξίας, σημασίας πολιτικής, να έχει κανείς σημαντικές ιδέες, σπουδαίες ιδέες για να πείσει το εκλογικό σώμα. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο ιδιαίτερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ευρύτερη συμμετοχή γυναικών. Πρώτα απ' όλα, δυσκολία στο να συνδυαστεί επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή. Και ακόμα, οι διαφορές οι αμοιβών στους μισθούς της αμοιβέ. Για αυτές τις τελευταίες αμοιβέ να σας πω ότι έχω κάτι το πολύ άσκημο σαν νέο Στη χώρα μου είναι μόνο 8% αυτή η διαφορά. Λιγότερο από το 16-17% στις υπόλοιπες χώρες. Αλλά σημαντικό να δώσουμε τη μάχη μας κατά αυτής της διαφοράς. Για το απλό γεγονό ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια αμοιβή από τη στιγμή που προσφέρουν την ίδια εργασία. Πολλά ιδιαίτερα ενδιαφέρθηκα ακούστηκαν κυρίως από την καθηγήτρια κυρία Ντάλερουπ, που φαίνεται ότι οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται τόσο να συμμετάσχουν σε εκλογές, τουλάχιστον σε σύγκριση με τους άνδρες. Και εκεί που υπάρχει ευρύτερη εκπροσώπηση γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, εκεί αντίθετα ενδιαφέρονται περισσότερο για τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να τους πούμε στις γυναίκες, να τους εξηγήσουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ποιο είναι το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παρνασχάρη, να είναι κάτι το σαφές, το διάφανο η εργασία αυτή, ώστε να ενδιαφερθούν και να πάνε και να ψηφίσουν και εκεί όπου εκπροσωπούνται λιγότερες γυναίκες στις χώρες αυτές και μέσω των νόμων για τις ευκαιρίες και για, με τις ποσοστώσεις προσέφεραν καλύτερα αποτελέσματα για υψηλότερη εκπροσώπηση γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά και για τη μάχη κατά της αποχής να πηγαίνουν οι γυναίκες να ψηφίζουν. Αυτό είναι το έργο μας, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες, όχι μόνο για το εκλέγεστε αλλά και για το εκλέγειν. Εντάξει, στις προσεχείς εκλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Αντιπρόεδρο. Τώρα θα μιλήσει Μία άλλη βουλευτής από την Πορτογαλία είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλο ιδιαίτερος την Επιτροπή Γυναικών που οργάνωσε αυτή τη διάσκεψη. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι οι εθνικοί εκπρόσωποι κάνουν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις ε, σε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι που βλέπω τόσες πολλές γυναίκες. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας. Είμαι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και ανήκω ε, και σε μια ε, υποεπιτροπή του, της Πορτογαλικής Βουλής για την, τα ίσα δικαιώματα στον οικογενειακό χώρο ανδρών και γυναικών. Ασχολούμαστε επίσης με θέματα μισθολογικής ε, αμοιβή, ε, με θέματα βίας κατά των γυναικών κτλ. Μετά από αυτά που είπε η συμπατριώτησά μου, ε, θα ήθελα εγώ να προσθέσω κάποια πράγματα. Πρόσφατα υιοθετήσαμε τον νόμο για την ισότητα. Στην πραγματικότητα μεταφέραμε ένα κανόνα που υπήρχε στο εσωτερικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος και υποβάλαμε αυτό το κείμενο προς στην Πορτογαλική Βουλή. Αυτός ο νόμος ισότητας προβλέπει ότι 33,3% ε, των εκπροσώπων θα πρέπει να είναι γυναίκες. Ελπίζω μέσα σε 10 χρόνια αυτός ο νόμος θα φτάσει στο να προστατεύει τους άνδρες. Ε, γιατί τα πράγματα θα έχουν αντιστραφεί. Αλλά σήμερα πρέπει να προστατεύσουμε τις ε, γυναίκες. Στην Πορτογαλία, με βάση τις ε, μελέτες, προκύπτει ότι βρισκόμαστε σε όλα τα επίπεδα κάτω από το 50% εκπροσώπηση και συμμετοχή των γυναικών. Επομένως, η μεγάλη πρόκληση είναι να υπάρχει παρουσία στους εκλογικούς καταλόγους των γυναικών, να εκλέγονται και οι γυναίκες, να εκλέγονται σε διευθυντικές θέσεις. Λέμε ότι μία θέση στις τρεις θα πρέπει να καταλαμβάνεται από γυναίκα. Ε, θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε οι γυναίκες να είναι ουραγοί σε όλα τα επίπεδα και ουραγοί στους εκλογικούς καταλόγους. Ελπίζω αυτό να ισχύσει σε όλα τα επίπεδα της χώρας μου, ε, στις τοπικές αρχές, περιφερειακές και εθνικές. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί ήδη υπάρχει μια τέτοια εκπροσώπηση. Σε ό,τι αφορά το τοπικό επίπεδο, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη υποεκπροσώπηση στην Πορτογαλία των γυναικών. Ελπίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο θα καλύψουμε τα κενά. Πρόεδρος, ευχαριστώ για όλα όσα μας είπατε. Θα ακούσουμε τώρα μια συνάδελφο από την Σλοβακία, την κυρία Πρεσίνσκα, η οποία επίσης είναι μέλος της Επιτροπής ε, γυναικών. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είστε εδώ, κύριε εκπρόσωπε της Τσεχικής Προεδρίας. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που συζητάμε σήμερα, τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που είχα τη δυνατότητα να δουλέψω επί πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Οι γυναίκες έδειξαν ότι πραγματικά μπορούν να παίξουν το δικό τους ρόλο στην πολιτική. Έχουν θέση, τη θέση τους ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία ισότιμα με τους άνδρες. Η δική μας Επιτροπή έχει στείλει πολύ θετικά μηνύματα και τα μηνύματα αυτά έχουν γίνει πράξη ε, και σε εθνικό επίπεδο, καλά προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πραγματικά έχουν επιβληθεί στο χώρο τους. Έχουμε υλοποιήσει μέτρα για να απλουστεύσουμε τις μικροπιστώσεις που δίδουμε σε γυναίκες. Θα πρέπει να πείσουμε τις γυναίκες να συμμετάσχουν στις εκλογές και μάλιστα να, πείσουμε όλους τους εκλογείς να προσφύγουν στις κάλπες. Οι γυναίκε θα πρέπει όμως να συμμετέχουν πολύ περισσότερο γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ακούσουμε και μια διαφορετική φωνή, μια διαφορετική άποψη. Και νομίζω ότι η σημερινή διάσκεψη πραγματικά θα μας βοηθήσει για να προχωρήσουμε, για να υλοποιήσουμε το στόχο μας του 50-50. Με αυτόν τον τρόπο Νομίζω θα βοηθηθούν και οι προεκλογικές εκστρατείες στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτός ο στόχος θα υλοποιείται σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν 10 γυναίκες στην, της ομάδας μου που συμμετείχαν στη σημερινή συνεδρίαση. Όλες αυτές οι γυναίκες νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν για να αλλάξουν τα πράγματα στη Σλοβακία. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε μία εκπρόσωπο της Κροατικής Βουλής, την κυρία Καρμέλα Καπαρίνα. Είναι μέλος της Επιτροπής των δικαιωμάτων των γυναικών. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για όλη την κοινωνία. Μόνο μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία υλοποιεί το δυναμικό της και δίνει στις γυναίκες τις θέσεις που τους ανήκουν. Τον Ιούλιο του 2008 το κοινοβούλιο μας υιοθέτησε ένα νόμο για την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών, ε, κυρίως μέσω της, των ποσοστώσεων για τα πολιτικά κόμματα. Ε, βέβαια, οι ποσοστώσεις είναι αμφιλεγόμενο θέμα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό εργαλείο για να αυξήσουν την πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Αυτή τη, στιγμή, η συμμετοχή των γυναικών επαφίεται στα χέρια των πολιτικών ηγετών. Με αυτόν τον τρόπο όμως ε, αναγνωρίζουμε ότι οι γυναίκες είναι πάνω το 50% του πληθυσμού της χώρας μας και ότι είναι α, εκ των όνου κάνευ για την ανάπτυξη της δημοκρατία, ε, δημοκρατίας καθώς και για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ γνωστό ότι συνήθως οι γυναίκες ε, βαραίνονται με μεγαλύτερο άχθος, ε, ειδικά σε κοινωνίες ε, που διανύουν περι, περιόδους κρίσης. Είναι λοιπόν δίκαιο ε, να δώσουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στις γυναίκες σε όλα τα όργανα και μηχανισμούς λήψης των αποφάσεων και στις διευθυντικές θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε έναν τρόπο επίσης να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες για να εμπλακούν πιο ενεργά στην πολιτική. Ε, ίσως αυτό είναι αρκετά δύσκολο για παραδοσιακούς και ιστορικούς λόγους. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια ε, και την κατάλληλη εκπαίδευση, τις κατάλληλες δημόσιες εκστρατείες, να ευαισθητοποιήσουμε τα ΜΜΕ, να, να προωθήσουμε συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και νόμους. Οι νόμοι βέβαια από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμοστούν. Επίσης, στις εκλογές που θα γίνουν ε, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα γίνει ε, μία πρώτη δοκιμή για το κατά πόσον θα συμπεριληφθούν περισσότερες γυναίκες υποψήφιες πάνω-πάνω στους εκλογικούς καταλόγους. Με βάση τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης συνεδρίασης ε, που έγινε στο, Ευρωπαϊκό, στο Κοινοβούλιο της Κροατίας, όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, συμφώνησαν ότι είναι η ώρα να συμμετάσχουν περισσότερο οι γυναίκες στην πολιτική και ότι αυτό θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Θα βοηθήσει πραγματικά την ευημερία της κοινωνίας μας εν το συνόλο της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα μπορούμε να ακούσουμε Την κυρία Κρέτου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, γνωρίζουμε ότι μερικές φορές ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν είναι και τόσο ευχαριστημένοι με την πολιτική και τους πολιτικούς. Τους πολιτικούς τους βλέπουν σαν άτομα που τους ενδιαφέρει εξουσία και όχι ο κόσμος ότι θέλουν να κρατήσουν την εξουσία αυτή. Εδώ δεν είναι ευχαριστημένος ο κόσμος αλλά από τη μία χώρα στην άλλη κυμαίνεται αυτό το ποσοστό έλλειψη ικανοποίησης. Η πολιτική μερικές φορές ε, είναι περισσότερο διεφθαρμένη και όχι δημόσια διοίκηση. Και όλα αυτά μας αποδεικνύουν κάτι. Εκεί που οι γυναίκες εκπροσωπούνται ευρύτερα οι δαπάνες για την υγεία, για την εκπαίδευση αλλάζουν, επαναλαμβάνω, λόγω αυτής της συμμετοχής, ενώ για την ναι, έμεινα, για την ασφάλεια, εξουσία, διάφορες υπηρεσίες ε, πληροφοριών κλπ. Αυτά τα έξοδα, αυτές οι δαπάνες είναι υψηλότερες αν υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες ε, και ακόμα για το ότι η ανάληψη κίνδυνου εξαρτάται και από το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών. Είναι σαφές ε, το μήνυμα, να μην πιστεύουμε όλα αυτά τα αραχνιασμένα πιστεύω τα παλιότερα. Οι γυναίκες έχουν την επαγγελματική πείρα, έχουν τα προσόντα το 57% των, όσων ε, ε, έχουν διπλώματα πανεπιστημίου είναι οι γυναίκες ε, το κούραγιο, η πολιτική βούληση. Τα διαθέτουν όλα αυτά οι γυναίκες. Κάτι άλλο δεν έχουν. Δεν έχουν χρήματα, δεν φαίνονται δημοσίως, γιατί σε πολλές χώρες έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Εκείνοι που έχουν την εξουσία φανίζονται περισσότερο στον τύπο, ε, μέτρα χρηματοδότησης, το ένα το άλλο. Ενώ οι γυναίκες όχι. Και κάτι ακόμα που μας λείπει είναι μια κατάλληλη οργάνωση δημόσιο χώρο για να εκφραστούν οι γυναίκες. Μερικές φορές μας λείπει και με ένα συνδυασμό ανάμεσα στην ζωή στην εργασία και στην ειδική ζωή και στα καθήκοντα στο σπίτι θα χρειάζεται μια πολιτική βούληση. Η ιστορία δεν είναι κάτι το φυσικό, είναι μεταρρυθμίσεις, είναι επαναστάσεις νομοθετικές και εμείς θα πρέπει να προσπαθήσουμε για αυτές τις μεταρρυθμίσεις νομοθετικές, για ίσες ευκαιρίες, για ίση εκπροσώπηση των γυναικών σαν πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέτου. Τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο η κυρία Μαργαρίτα Πέτκοβα από τη Βουλγαρία. Добър ден на всички. Голямо удоволствие за мен да направя едно малко уточнение, че... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά έρχομαι για να μιλήσω εδώ και να κάνω την εξή μικρή διευκρίνηση. Οι γυναίκε οι οποίε δραστηριοποιούνται στην πολιτική στη Βουλγαρία την χάνουν εκτίμηση όχι μόνο για τις καμπύλες τους, αλλά για το ρόλο τους και τις δραστηριότητες τους στην πολιτική μας ζωή και αποτελούν υπερηφάνεια, λόγω υπερηφάνειας για μας όλους τους Βούλγαρους. Χαίρομαι λοιπόν για την ευκαιρία που μας δόθηκε με αυτή τη διάσκεψη. Συγχαίρω τους συνεργοδοτές της και υπενθυμίζω ότι σήμερα και κατά τη διάρκεια των ερωτασμών ε, της, ημέρας, ε, της ημέρας της Γυναίκας εμείς εκπρόσωποι των οργανώσεων των σοσιαλιστριών γυναικών κάνουμε και από το δικό μας μετερίζει ό,τι μπορούμε για να ε, καταπολεμήσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα δεινά της οικονομικής κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Και για μια φορά, καλή ημέρα της γυναίκας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Επίσης και από εμάς τις καλύτερες ευχές. Και τώρα μπορώ να δώσω το λόγο στην κυρία Παγκάνο βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του συναδελφού μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εντύπωσή μου είναι ότι οι διεθνή θέματα άλλαξαν με κέντρο ενδιαφέροντος λόγω ακριβώς της κρίσης που επιδεινώνει τις συνθήκες ζωής των πολιτών, κυρίως εις βάρος των γυναικών. Το κοινωνικό θέμα είναι ησυχία για την εργασία. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητα και εκπροσώπηση έτσι ίσως γίνει δευτερεύουσα σημασίας που είναι για ορισμένες μικροελίτ πολιτιστή που ασχολούνται με παρόμοια πολιτιστικά στα πούμε θέματα και στην Ιταλία φτάσαμε στα 540% στο Ταμείο Ανεργίας και 21% ανεργία στο Νότο και πολλές ε, με διπλώματα πανεπιστημιακά ή ανώτερα διπλώματα και τα μεσαία στρώματα επίσης γίνονται πιο φτωχά και όλα αυτά ε, κλέβουν τον ρόλο σημασίας από αυτά που εμείς συζητούμε και απομακρύνουν τις γυναίκες από την πολιτική κούραση η πολιτική και τώρα περικόπτουν υπηρεσίες και δυνατότητες εξεργασίας για τις γυναίκες και ο χρόνος είναι όλο και λιγότερος για να ασχοληθεί κανείς με να δώσει πολιτικές μάχες. Αλλά η παρουσία όπως υπόθηκε εδώ για τις γυναίκες ε, είναι κάτι το βασικό για να αλλάξει η κοινωνία. Σίγουρα η εκπροσώπηση από εκεί εξαρτάται και το κίνημα των γυναικών ε, στις χώρες από τις οποίες προερχόμαστε και χθες σαν Ευρωβουλευτές ακούσαμε και τη μαρτυρία του βραβείου Νόμπελ για την ειρήνη από το Ιράν που είπε η κυρία αυτή ότι το κίνημα των γυναικών στο Ιράν είναι πολύ ισχυρό που κάθε φορά που κάποιος φυλακίζεται δίνεται ιδιαίτερη μάχη για να αποφυλακιστεί. Και είναι σημαντικό το κίνημα αυτών των γυναικών, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο γυναικών. Όπως είπε όμως και η καθηγήτρια που είπε προηγουμένως, όλα αυτά σχέση και με, έχουν σχέση και με τα εκλογικά συστήματα. Αναλογικό, καθαρό αναλογικό σύστημα όπως οι ευρωεκλογέ, ας πούμε στην Ιταλία Εκεί μετράμε τις ψήφους προτίμησης ε, και απαιτούνται 120.000 ψήφοι για την εκλογή στο Κοινοβούλιο και το 50% των γυναικών να πάνε σε ένα ρόλιο ψηφοδέλτιο ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει κίνδυνο να μην εκλεγεί ούτε μία γυναίκα. Αυτό το σύστημα έχει τρομερή σημασία. Η καθηγήτρια που μίλησε προηγουμένω έχει δίκιο που το υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προσφέρουμε και ενδείξει όσον αφορά τα τα εθνικά συστήματα σε σχέση τουλάχιστον με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακόμα για τις οικονομικές κυρώσεις. Δεν φτάνουν αυτές. Γιατί εκεί αυτό που ισχύει είναι ότι εμεί όπω πριν από κάποιο χρονικό διάστημα στην Ιταλία, στο Κοινοβούλιο, είχαμε μια οικονομική κύρωση για τα ψηφοδέλτια που δεν συμπεριλάμβανε γυναίκε. και πολλά κόμματα προτίμησαν να ψηφίσουν αυτό το, να πληρώσουν αυτό το πρόστιμο παρά συμπεριλάβουν γυναίκε που θα εκλεγούν. Άρα λοιπόν η μοναδική κύρωση είναι να μην μπορεί κανεί να κατεβάσει υποψηφίου ε, σε ψηφοδέλτια από τη στιγμή που δεν υπάρχει το απαραίτητο ποσοστό γυναικών. Αυτό είναι το πρόβλημα και πώς θα πρέπει να, αντιμετωπίσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ιακωβή παρακαλώ, μπορεί να λάβει το λόγο από το Κοινοβούλιο της Μακεδονίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μεγάλη χαρά που προστάνομαι σήμερα που είμαι εδώ κοντά σα, θέλω να σα πω μερικά λόγια για τι γυναίκε στη χώρα μου, τη Μακεδονία. Είμαι βουλευτής δημοκρατική του κόμματος, του Δημοκρατικού Κόμματος της ε, ε, ενσωμάτωσης αλβανόφωνου κόμματος με οκτώ γυναίκες στο Κοινοβούλιο. Εμείς στη Μακεδονία έχουμε 32% εκπροσώπηση των γυναικών στο κοινοβούλιο μας. Με συγχωρείτε για τα αγγλικά μου λέει η ομιλήτρια, δεν ε, τα κατέχω τόσο καλά. Θα ήθελα να μιλήσω αν μου επιτρέπετε μακεδονίτικα και να μεταφράσει συνάδελφος δίπλα μου.

και έχουμε 29 βουλευτές στο κοινοβούλιο της χώρας, εκ των οποίων 8 είναι γυναίκες. Αντιστοιχεία δηλαδή, ε, αναλογία δηλαδή 27% των δικών μας βουλευτών, ε, των αβανόφωνων, είναι γυναίκες στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Στο κόμμα μου γυναίκες βουλευτές είχαμε και πριν από την εισαγωγή του συστήματος των ποσοστώσεων υπέρ των γυναικών. με χαρά διαπιστώνουμε ότι στη χώρα μου και ότι έχουμε ποσόστοση κατά 30, για, για αναλογία 30% των γυναικών εκ του νόμου. Έχουμε υπερβεί το ποσοστό αυτό και τώρα έχουμε αγγίξει το 32% συμμετοχή των γυναικών στο κοινοβούλιο. Μέχρι τις παρούσεις είχαμε τρία διαφορετικά πρότυπα ε, ποσοστώσεων, τρία διαφορετικά συστήματα ποσοστώσεων στη χώρα μου. Για πρώτη φορά το 2002 είχαμε ένα, ποσοστό, ένα σύστημα ποσόστοσης με ποσοστό 30% των γυναικών στον εκλογικό κατάλογο, στη λίστα δηλαδή, με αποτέλεσμα όμως συμμετοχή 8,3 μόνο των γυναικών στο Εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί το 30% των γυναικών δεν εκπροσωπήθηκε σε υψηλέ θέσει ή εκλόγιμες και ήταν μάλλον προς το τέλο τη εκλογική λίστα. Γι' αυτό δεν με αρκετέ γυναίκε. Τη δεύτερη φορά, το δεύτερο σύστημα, το είδαμε στι τελευταίε τοπικέ εκλογέ πριν από τέσσερα χρόνια με μία ποσόστοση για 30% των γυναικών στο άνω ίμιση της λίστας και άλλο 30% στο κάτω ίμιση με αποτέλεσμα μια αρκετά καλή εκπροσώπηση των γυναικών στις δημοτικές λίστες. Και τώρα, την τελευταία φορά του 2006 για τις κοινοβουλευτικές εκλογές, είδαμε ότι μπορούσαμε να έχουμε για τους τρεις πρώτους υποψηφίους ε, εναλλαγή φύλων με το νέο σύστημα και έτσι στις τελευταίες εκλογές το 2008 είδαμε ότι μπορούσαμε να αγγίξουμε το 31% 31,7% ε, συμμετοχή των γυναικών στο Εθνικό Κοινοβούλιο με αποτέλεσμα ότι ένα πολιτικό κόμμα μπόρεσε να δείξει εμπιστοσύνη στις γυναίκες και να βάλει ακόμη περισσότερες γυναίκες από όσες το υποχρέωνε ο νόμος στο η λίστα. Εγώ είμαι βουλευτής ε, στην Επιτροπή που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, για τις ευκαιρίες. Αγωνίζομαι και για, τις τοπικές, ε, για την τοπική δράση και για τις τοπικές εκλογές, για περισσότερη εκπροσώπηση δηλαδή, των γυναικών, γιατί τώρα μόλις αρχίζει αυτή η μετάλλαξη στην ε, χώρα μου. Και έτσι ελπίζω ότι με τις προσεχείς τοπικές εκλογές θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ε, παρουσία των γυναικών. Από το 22,7% ελπίζουμε ότι θα πάμε στο 30% και περισσότερο. Ότι θα καλυφθεί η ποσόστοση αυτή και ελπίζουμε μια μέρα να δούμε γυναίκα πρόεδρο Κοινοβουλίου του Κοινοβουλίου μας. Αν και πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε αντιπροέδρους, δύο τουλάχιστον ε, γνωρίσεις στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Στην Επιτροπή μου επίσης αγωνιζόμαστε για να εξασφαλίσουμε περισσότερη, ε, εντολότερη μάλλον παρουσία γυναικών στις, ε, στους ανώτερες θέσεις, διαχειριστικές κύριες θέσεις, σε κάθε τομέα δραστηριότητας της κοινωνίας μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο η κυρία Φρανσέσκα Μελίνα που εκπροσωπεί το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από δική μας πλευράς, από την προσωπία μας, από το ε, Ισπανικό Κοινοβούλιο, τιμή μας που είμαστε εδώ να σας δώσουμε συγχαρτήρια και στην Επιτροπή σας για την οργάνωση αυτής της σημερίδας να εκφράσω ορισμένες σκέψεις και απόψεις σχετικά με το θέμα που σήμερα το πρωί συζητάμε εδώ. Να υπογραμμίσω τη σημασία να έχει κανείς νομοθετικά μέσα νόμους, ώστε να μπορέσουμε να δούμε από πού προέρχεται αυτή η λήψη ισότητας. Είναι... Είμαστε πρωτοπόροι εμείς στη χώρα μας, στην Ισπανία, για τα νομοθετικά μέσα νόμος ισότητας ή κατά της βίας εις γυναικών. Και σε αυτή την κρίση την οικονομική που ζούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήθελα να πω ότι αυτό το σύστημα είναι ανεπαρκές γιατί διατηρεί πολλά προβλήματα ανισότητας των δύο φύλων. Χρειάζεται ένα νέο πρότυπο ισότητας να είναι υπεύθυνοι και οι δύο, είναι υπεύθυνοι άνδρες και γυναίκες με μια σημαντική ψυχή και δεν θα πρέπει να πεισοδρομήσουμε σε όσα δικαιώματα είναι δικαικτημένα. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε βέβαια, αλλά ταυτόχρονα να παγιώσουμε ορισμένα που ισχύουν. Ε, αυτό αποτελεί το στόχο της εργασίας μας, την πρόκλησή μας, τα προσεχή έτη και θα προσεχείς επίσης ευρω... εκλογές. Σας ευχαριστώ. E, ευχαριστώ πολύ την εκπρόσωπο του Ισπανικού Κοινοβουλίου και πριν δώσω το λόγο στην προσοχή ομιλητή ή ομιλήτρια, θα ήθελα να κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε ακόμη να ακούσουμε τρεις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο η κυρία Μύρια Μπάσκη, Γενική Γραμματέας του Λόπι των Γυναικών. Καλημέρα. Δυστυχώ η Γενική Γραμματέα μα ε, χρειάστηκε να φύγει εσπερισμένο γιατί είχε ένα προσωπικό πρόβλημα. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρου τη. Θα μιλήσω εξ ονόματό τη. Ε, από το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών που εκπροσωπούν περίπου 2.000 οργανώσει. Ε, 2.000 οργανώσει είναι μέλη του Λόμπι και 30 ε, ευρωπαϊκοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Η εκστρατεία μα για τη δημοκρατία έχει σαν σκοπό να εκπροσωπήσει ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα εκλεγού, κοινοβούλιο που θα εκλεγεί από τις επόμενες εκλογές του Ιουνίου του 2009. Ε, υπάρχουν ε, προσωπικότητες που συμμετέχουν ε, από την Ευρώπη, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία ε, Βάλστρομ, η Ντένιλο Τούρκ, από τη Σλοβενία, το, ο Ορκάν Παμούκα, βραβείο λογοτεχνίας, ο Ερμαν Βάλτεν Χόι, ε, και ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σιμών Βέιλ. Ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2008 αυτή η εκστρατεία και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2009, δηλαδή μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές και μέχρι το διορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εκστρατεία αυτή ε, προβλέπει εκδηλώσει όλη την Ευρώπη. Για να υπάρξει μια δίκαιη δημοκρατία θα πρέπει να εκπροσωπηθούν όλες οι Ευρωπαίες και Ευρωπαίοι, γυναίκες και άνδρες, στη λήψη των αποφάσεων, ε, αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Η εκπροσώπηση λέει ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψη των αποφάσεων στην Ευρώπη ε, οδηγεί στην έλλειψη δημοκρατικής νομιμότητας της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, πολλές δεσμεύσεις ελήφθησαν για τη δημοκρατία και την ισότητα ε, και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Το 77% ε, των μελών του Κοινοβουλίου ε, είναι άνδρες και το 66% των επιτρόπων είναι άνδρες. καλούμε τους εκλογές άνδρες και γυναίκες, τις, τους υπεύθυνους, τους ηθήνοντες των πολιτικών κομμάτων, τα πολιτικά κόμματα να δράσουν ούτω ώστε αυτή η απεικόνηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας στα πολιτικά όργανα να είναι πιο ισότιμη υπέρ των ανδρών και υπέρ των γυναικών. Έχουμε μια εκπρόσωπο του European Disability Fund. Παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ λοιπόν το ε, European Disability Forum το οποίο εκπροσωπεί τι οργανώσεις ε, ανθρωπιστικές που ασχολούνται με τους ανθρώπους με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί στασόμαστε 100% υπέρ της ε, ποσόστοσης της εκστρατεια 50 50-50. Και θα ήθελα να σα δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε 50 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίε στην Ευρώπη, εκ των οποίων 55 με 60% είναι γυναίκε γυναίκες με αναπηρία. Ε, στο θέμα λοιπόν των διακρίσεων, οι γυναίκε με αναπηρίες έχουν πέσει όλο και περισσότερο, είναι θύματα πολύ περισσότερο μια αρνητική ε, διάκριση από ότι ένα άντρα με αναπηρία ή μια γυναίκα χωρί αναπηρία. Επίση, μια γυναίκα με αναπηρία έχει συχνά εμπλοκή και ανάμειξη στον πολιτικό βίο, στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Με την εκστρατεία για τις ευρωεκλογές του 2009 λοιπόν, αλλά και με την ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας της γυναίκας, δημοσιεύσαμε ένα μανιφέστο για τα δικαιώματα των γυναικών, μάλλον για τα δικαιώματα των φίλων και την ισότητα των φίλων με δέκα κύριε απαιτήσει και διεκδικήσει. σε μία όμω θα αναφερθώ μόνο που σχετίζεται και με το σημερινό θέμα μας. Το δικαίωμα δηλαδή για ισότιμη πρόσβαση στι ε, προεκλογικέ εκστρατείε και τι εκλογικέ αναμετρήσει, Το δικαίωμα του εκλέγει ω θεμελιώδε δικαίωμα και εκλέγει με μία πλήρη και περιστατωμένη ενημέρωση για τους υποψηφίους. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πρόσβαση σε πληροφορία κατάλληλη, επί παραδείγματι σε μπράιλ, σε ε, νοηματική γλώσσα, όπως άλλωστε ακούσαμε και νωρίτερα σήμερα, σε υποτιτλισμό των προγραμμάτων της τηλεόρασης, όταν πρόκειται για ε, προεκλογικές συζητήσεις ή αναμετάδοση και ηχητική ορισμένων εικόνων της τηλεόρασης ώστε να μπορεί να παρακολουθεί ε, κάποιος που έχει προβλήματα όρασης. ισότιμη πρόσβαση επίσης στην προεκλογική εκστρατεία σημαίνει και δικαίωμα του εκλέγεσθε και ενθαρρύνουμε γυναίκες με, τη, με αναπηρίες, πιστεύω θα πρέπει γυναίκες με αναπηρίες να ενθαρρύνονται να υψώνουν το ανάστημα και να συμμετέχουν στι εκλογικέ αναπετρήσει. Το μανιφέστο μα. το βλέπετε εδώ, το έχουμε αφήσει στο τραπέζι στο πίσω μέρο τη αίθουσα. Παρακαλώ όποιο ενδιαφέρεται να πάρει αντίγραφα και θα ήθελα να σα ενημερώσω επίση και για την ιστοσελίδα μα εν ώψη των ευρωεκλογών που έχει το όνομα Disability Votes Count γιατί πιστεύουμε ότι 50, εκατομμύρια ανθρώπων με αναπηρίες, εκ των οποίων περισσότερο από το μισό είναι γυναίκες, είναι ψήφοι που μπορούν να φέρουν πολύ μεγάλη διαφορά, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό λέμε disability votes count. Οι ψήφοι της αναπηρίας μετράνε, υπολογίζονται. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ την κυρία Ειρήνη Παπάντσεβακ από την Βουλγαρία να λάβει το λόγο. Εκπροσωπεί επίση το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για άτομα με αναπηρίες. Παρακαλώ. Okay, uh, thank you very much. Ευχαριστώ η συνάδελφός μου, η Βαλερή, εξέφρασε τις προσπάθειες που κάνουμε, τις ανησυχίες που έχουμε. Ε, δουλεύω και εγώ για το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Και θα ήθελα πραγματικά να υποστηρίξω θερμά και να προσυπογράψω τα λόγια της. και να κάνω έκκληση. να συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες στην πολιτική και μάλιστα περισσότερες γυναίκες με αναπηρίες στην πολιτική. Ευχαριστώ. Στη συζήτηση αυτή έλαβαν μέρο πολλοί άνδρε και πολλέ γυναίκε. Ακούστηκαν πολλές απόψει. Έχουμε σχεδόν φτάσει στο τέλος της συνεδρίασή μας. Και επιτρέψτε μου τώρα κλείνοντα και κλείσοντας το τέλος των εργασιών μας να πω δύο λόγια συμπερασματικά. Βλέπουμε ότι επαναλαμβάνονται τα προβλήματα ότι έχουμε πάντα την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο φύλων και τα κύρια προβλήματα παραμένουν δυστυχώς τα ίδια. Πιστεύω πάντως ότι έστω και με κάποιους αργούς ρυθμούς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ε, πρόοδος, ότι έχει βελτιωθεί η θέση, ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία μας σήμερα. Ο Επίτροπος και η κυρία Επίτροπος αναφέρθηκε σαν σε ορισμένα αριθμητικά στοιχεία που με κατέπληξαν δηλαδή το πρόβλημα της ε, διαφοράς που ανέφερε ο κύριος Σπίγκλα μεταξύ των αμοιβών που προσφέρονται σε άνδρες και γυναίκες για την ίδια δουλειά. φωτόθηξε και η κυρία Βάλστον βέβαια. Ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει οξυμένο. Επίσης, Το θέμα αυτό για πρώτη φορά, αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, πριν από 52 χρόνια εισήχθη ως στοιχείο και διεκδίκηση του της ευρωπαϊκής κοινότητας τότε με τη συνθήκη της Ρώμης του 1957 όπου γινόταν λόγος για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών ή καλύτερα για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και ακόμη μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, 52 χρόνια μετά, δεν φτάσαμε στην ίση αμοιβή. Και εδώ πάλι δεν μπορούμε να αποδώσουμε τις ευθύνες αποκριστικά στην νομοθεσία. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη καλής βούλησης, η, η παραδοσιακή θέση της ε, γυναίκας στην κοινωνία, θέματα που έχουν να κάνουν και με τη φτώχεια και με τη βία και με το εμπόριο ανθρώπων και με την ε, ε δυναμία αναρρίχησης γυναικών σε αποφασιστικές ε, κρίσιμες θέσεις στην ηγεσία των επιχειρήσεων της πολιτικής. Και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι μπορεί η αρχή της ε, ισότητας ή καλύτερα της δικαιοσύνης θα αρκούσε για να λυθούν πολλά από τα προβλήματα. Εάν κρίναμε δηλαδή τα πράγματα μόνο με γνώμονα την δίκαιη, την ισότιμη μεταχείριση. Αυτό είχα να προσθέσω μόνο εγώ συμπερασματικά. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ. Πάνω από όλα χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθαν τόσοι πολλοί εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων και πριν ε, κλείσω το μικρόφωνο θα ήθελα να απευθύνω προς όλους ε, τους και τις εδώ παρούσες και παρόντες, όχι μόνο ε, άνδρες ή γυναίκες πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για όλους όσους μας ακούνε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να απευθύνω λοιπόν τις καλύτερες ευχές για την Εθνή μέρα της γυναίκας και πάνω απ' όλα την ευχή να αξιοποιεί ο καθένας όποια ευκαιρία του προσφέρει η κοινωνία του για να προχωρεί και βέβαια για το καλό όλων, για να προχωρεί η κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές που είχαμε εδώ στο πάνελ, όλους τους ε, βουλευτές και τις βουλευτές που ήταν εδώ και που μίλησαν. Ευχαριστώ τη Γραμματεία της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της ε, Ισότητας Μεταχείρισης των Φίλων των Δικαιωμάτων και βέβαια το προσωπικό που μας ε, ε, υπηρετεί πάντοτε στις ε, συνεδριάσεις μας. Ευχαριστώ τους Γερμηνείς, λέει πολύ ευγενικά η Πρόεδρος, οι οποίοι μας, οι οποίοι μας επέτρεψαν να συνεννοηθούμε σε αυτή την πολύγλωση κοινωνία. Ευχαριστούν και οι Διερμηνείς από την πλευρά τους. Και ήθελα, κλείνοντας, να σας προσκαλέσω όλες και όλους σε μια δεξίωση που θα λάβει χώρα εδώ, στο κτίριό μας, Φεύγοντας λοιπόν από την ε, αίθουσα στην οποία βρισκόμαστε, δεν χρειάζεται παρά να κατέβετε έναν όροφο πιο κάτω, στο δεύτερο όροφο, στο κτίριο που ονομάζεται Atrium, πάλι εδώ δηλαδή, για να ε, συμμετάσχετε και εσείς στη δεξίωση. Ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι θα είναι πολύ μεγάλη η επιτυχία των γυναικών και της κοινωνίας μας γενικότερα στις προσεχείς ευρωεκλογές ešte, eh, ak dovolíte jednu... Δεν μπορούμε βέβαια να αφήσουμε τη μεγάλη ευκαιρία όπως η σημερινή συνάντηση να μείνει χωρίς κάποιο αναμνηστικό. Μας περιμένει ο φωτογράφος λοιπόν εδώ μπροστά από την αίθουσα.